Good day. Good day, everybody. Good day, everybody. Καλημέρα σας όλοι και όλες. Κυρίες και κύριοι, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι στην ακρόαση που οργανώνεται από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ. Σας πω Ποιος είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών και για μένα είναι τιμή που κηρύσω την έναρξη της ακρόασης αυτής που οργάνωσε ο εισηγητής μας κύριος Κορνέλης Ντε για το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο ή μάλλον για την ευρωπαϊκή αντίληψη του ποινικού δικαίου. understanding of the area of liberty. Γιατί ο χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας σημαίνει ότι πρέπει να ορίσουμε και την ευρωπαϊκή αυτή προσέγγιση του ποινικού δικαίου. Ξέρουμε ότι όταν τέθηκε ενισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας το Δεκέμβριο του 9. η ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια δεν ήταν πια αποκλειστικό αντικείμενο διακυβερνητικών συνεννοήσεων μεταξύ των χωρών μελών, αλλά επιτέλους κατέστη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Και άρα υπόκειται στη συνήθι νομοθετική διαδικασία που λέγεται συναπόφαση Για μας λοιπόν έγινε πολύ σημαντικότερο από ό,τι πριν να εκλισαβωνώσουμε αυτό το θέμα του πρώην τρίτου πυλώνα για να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων και ακόμα σημαντικότερο δικαστική συνεργασία όχι μόνο σε αστικά θέματα αλλά και σε ποινικά με συνεργασία αστυνομιών και διακαστικών αρχών όπως και κοινή αντίληψη για τα διαμεθοριακά σοβαρά εγκλήματα. Έτσι τα άρθρα 67 με 89 το προβλέπουν και έτσι σκοπεύει και η Επιτροπή μας να προωθήσει το θέμα. Μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια έχει οργανώσει πολλές συζητήσεις του. Γι' αυτό και εγώ τονίζω τη σημασία της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας που έχει συγγράψει ο κύριος Κορνίλης Ντεχιόγκ που θα προεδρεύσει στη συνέχεια των διαδικασιών εδώ και θα κάνει την πρώτη εισήγηση και θα μας παρουσιάσει και τους καθηγητάς που έχουν προσκληθεί εδώ να μας κάνουν τις παρουσιάσεις τους για τις διάφορες πετυχές της ευρωπαϊκής αυτής προσέγγισης στο ποινικό δίκαιο σύμφωνα με την ομολογία που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε και εμείς χρήσιμα μία όντως ευρωπαϊκή προσέγγιση του ποινικού δικαίου. Εγώ θεωρώ ότι τα διαμεθοριακά εγκλήματα είναι από τις σημαντικότερες πτυχές της παγκοσμιοποίησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να το να απασχοληθεί και με αυτό. Τα διαμεθοριακά εγκλήματα είναι διεθνοποιήθηκαν πριν ακόμη τα υπόλοιπα. παγκοσμιοποίηση έδωσε και περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες αγορές, χρηματοδότηση, αλλά τα δικαιώματα και ιδίως το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια δεν παγκοσμιοποιήθηκαν επαρκώς. Υπάρχουν απειλές προς την ασφάλεια των όντων και πολιτών. και οι πολιτικοί παράγοντες δεν το αναγνώρισαν επαρκώς. Καθήκον μας είναι λοιπόν τώρα να το καταλάβουμε και να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει για να χορηγήσει πράγματι, να δημιουργήσει πράγματι τον χώρο ασφαλείας και ελευθερίας. Γι' αυτό και εγώ ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου έχω τονίσει ανέκαθεν. την υποδειγματική σημασία που έχει αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς η πτυχή του ενωσιακού συνταγματική της ενωσιακής συνταγματικής τάξης που μας προμήθευσε η Λισαβόν. είναι πολύ σημαντική έκφραση της συνταγματικής τάξης και αυτό, διότι το ποινικό δίκαιο έχει επιπτώσεις στην στην ομολογία των χωρών μελών. Η συνθήκη της Λισαβόνας έδειξε ότι και σε αυτό πρέπει να θέσουμε σε σε κοινή, να συμμετάσχουμε όλοι μαζί και στα αποτελέσματα της καταπολέμησης του διαμεθοριακού διεθνούς δηλαδή εγκλήματος, να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για την επιβολή του νόμου και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή η οργάνωση της ακρόασης. Προσδοκούμε με αδημονία στις συζητήσεις που θα γίνουν και συγχαίρω ακόμη μία φορά τον κύριο Κορνέλης Ντεγιόγκ που ανέλαβε είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που, που λέγω δέχτηκε και η Επιτροπή μας και φυσικά θα παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια που θα δοθεί, πώς θα μεταφραστούν δηλαδή οι προσπάθειες αυτές σε νομοθεσία και μάλιστα αποτελεσματική νομοθεσία για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο μας θα αφήσουμε βέβαια χρόνο για σχόλια και συζήτηση μετά από κάθε παρέμβαση των καθηγητών και προτείνω όποιος θέλει να πει κάτι ή να θέσει κάποιο ερώτημα να μην ξεχνάει ότι υπάρχει χρονικό περιορισμός. Όσοι θέλουν να μιλήσουν λοιπόν να περιοριστούν σε 2-3 λεπτά το πολύ ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε όλους και όλες Τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Κορνίλης Ντε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τα ευγενικά σας λόγια. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί τα υπόλοιπα όργανα έχουν εκπονήσει γνωμοδότηση για το πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ποινικό δίκαιο έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2009. Έχουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε πιο πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, έχει ακόμη εκπονήσει έκθεση για το θέμα αυτό. Έχουμε μία έκθεση για το οικονομικό ε, δίκαιο, αλλά για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο είναι ένα σχετικά νέο τομέα, ακόμη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και αν ε, κάποια λίγα μέτρα έχουν ήδη υιοθετηθεί αναπερίπτωση. Και καθώς ε, πρόκειται για ακρόαση, δεν θα με κρηγορήσω στην εισαγωγή μου. Νομίζω ότι θα ήταν ε, καλύτερο και ο εισηγητής ε, να ακούσει τους διακεκριμένους καλεσμένους που έχουμε σήμερα εδώ. Έχουμε αρκετούς και νομίζω ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν πολύ σημαντικά. Θέλω να πω ότι η ακρόαση προκύπτει και από την ε, δομή της εκθεσής μου. Ξεκινάμε με, την, ε, με το πρώτο θέμα και λέμε ας υποθέσουμε ότι υπάρχει περιθώριο για ποινικό δίκαιο, αλλά θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο μπλοκ της συζήτηση, το πρώτο τμήμα και για το δεύτερο τμήμα συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να έχουμε ποινικό δίκαιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποια είναι τα ορθά κριτήρια, τα ποιοτικά κριτήρια. Και στο τρίτο τμήμα έχουμε ένα πλαίσιο Ας ελπίσουμε, γνωρίζουμε τα κριτήρια, ότι θα υπάρχει νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια της καλής νομοθεσίας, καλής ποιότητας νομοθεσίας και το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούμε σε διοργανικό επίπεδο και είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι μπορεί να φαίνεται αρχικά γιατί σε εθνικό επίπεδο συχνά έχουμε το εξή σύστημα. Μπορεί να έχουμε ένα Υπουργείο Αρμόδιο, συνήθω το Υπουργείο Δικαιοσύνη, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα του ποινικού δικαίου εν γέννη. Και αυτό δεν έχει σημασία αν ε, μιλάμε για τον περιβαλλοντικό τομέα ή αν ε, μιλάμε για συμμετοχή παραδείγματος χάρη του Υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωση απάτης. Δεν έχει σημασία ποιο υποβάλλει την πρόταση. Πάντοτε θα υπάρχει τελικά ε, έλεγχο για την ποιότητα τη νομοθεσία από την κυβέρνηση. ακόμη και σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να υπάρχει γραφειοκρατία, αλλά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Α ε, δούμε αυτό το κοινοβούλιο, ω ε, παράδειγμα. Έχουμε πάρα πολλέ επιτροπέ ε, που όλε ασχολούνται και λίγο με το ποινικό δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει ε, κάπου που να συγκεντρώνονται όλα αυτά σε αυτόν τον οίκο. Κάποιο δηλαδή να ελέγχει αν οι ποινέ συνάδουν ε, μεταξύ τους ε, ή αν η περιγραφή των ε, αδικημάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο που να έχει νόημα αν συγκρίνουμε την περιγραφή άλλων αδικημάτων. Για να επανέλθω στο πρώτο θέμα, για το αν θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε. Στο ότι υπάρχει ήδη στη συνθήκη, παραδείγματο χάρη. Μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει ένα κατάλογο αδικημαντών στο άρθρο 83 παράγραφο 1 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. που αναφέρεται ρητά. Αυτά τα δικήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση. Αυτό είναι το ένα κριτήριο λοιπόν θα έλεγα. Έχουμε τον κατάλογο των αδικημάτων, έχουμε και ένα πρόσθετο κριτήριο που θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και άλλα αντικείμενα που δεν έχουν αναφερθεί ρητός ε, στη συνθήκη. Και έχουμε και τη δεύτερη δυνατότητα, ένα δίκημα να είναι ουσιαστικό για να διασφαλίσουμε την ε, ουσιαστική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης σε ένα τομέα που ήδη έχει τύχει μέτρων εναρμόνισης. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ήδη ένα είδος εναρμόνισης και το ποινικό δίκαιο στη συνέχεια είναι ουσιαστικό για να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι ανοιχτό ακόμη προ τη ζήτηση γιατί δεν υπάρχει συμπληρωθεί στη συνθήκη και δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην πράξη νομίζω, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια συζήτηση για το τι σημαίνει και ποια κριτήρια θα μπορούσαν να προσθεθούν. Και θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί είδαμε στην ανακοίνωση της Κομισιόν ότι περιλαμβάνονται και άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να, να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα. Η ιδέα, παραδείγματο χάρη, του Φόρουμ shopping από του εγκληματίε. Αν, παραδείγματο χάρη, ορίζονται διαφορετικά τα δικήματα στα διάφορα κράτη-μέλη, ενδιαφέρουν οι ποινέ, τότε θα μπορούσαν οι εγκληματίε ε, να πάνε εκεί όπου είναι σχετικά εύκολο ε, να διαπράξουν το έγκλημα ή παίρνουν το σχάρι, έχουν ε, πιο χαμηλή ποινή. Θα ακούσουμε τι θα μας πούν και οι ακαδημαϊκοί. Νομίζω ότι είναι κάπως αόριστο κριτήριο. Δεν βλέπω να υπάρχουν αποδείξεις και εξαρτάται πολύ ε, από το είδος του δικήματος. Νομίζω ότι απλή κλοπή Παραδείγματο χάρη διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά α ακούσουμε τους εμπειρογνώμονε Είναι νομίζω ένα θέμα προσυζήτηση. Και το δεύτερο σημείο, στο πρώτο τμήμα, είναι η αρχή της αναλογικότητας. Ε, αν έχουμε την επικορικότητα, έχουμε και την αναλογικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ποινικό δίκαιο. Γιατί πάντοτε διακυβεύονται ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή αφαιρούμε την ελευθερία κάποιου, ποινικοποιούμε κάτι και πρέπει να υπάρχει ένας νόμιμος ε, σκοπός. Και νομίζω ότι αυτό επίσης σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ζημία στην κοινωνία, βλάβη στην κοινωνία. Και επίσης έχουμε και την αρχή του ultima ratio, και όλα τα άλλα μέτρα που δεν συμπεριλαμβάνουν στοιχεία ποινικού δικαίου, δηλαδή δεν έχουν επαρκές αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ιδίω πολιτικοί όπως εμείς, δεν ασχοληθούν με αυτό, γιατί εγώ είδα επίση στι Βρυξέλλε ότι μερικέ φορέ στι εφημερίδε ε, υπάρχει κατακραυγή το χάρη και τι μπορεί να κάνει κάποιο ως πολιτικό. Στην ε, πιο εύκολη περίπτωση είναι να πει κάποιο ναι, είναι τόσο τρομερό που πρέπει να ποινικοποιήσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να προτείνουμε ε, νέες ε, ποινικέ κυρώσει. Αυτή είναι στερεότυπη αντίδραση πολιτικού σε ένα γεγονό, σε ένα συμβάν. Και ακριβώς αυτό που ισούν νομικοί γενικά. Γιατί δεν καθιστά σαφέ ότι έχουμε την αρχή ultima ότι είναι ο μόνος τρόπος δηλαδή να δημιουργήσουμε αυτό. Και αν αυτοί οι πολιτικοί που αντέδρασαν σε όσα λέγονταν στην εφημερίδα, δηλαδή είχαν σκεφτεί ποια με άλλα μέτρα θα μπορούσαν να πετύχουν το ίδιο στόχο, καλύτερο αυτό είναι λοιπόν το πρώτο τμήμα τη συζήτηση. Το δεύτερο τμήμα αφορά κυρίως τις αρχές που πρέπει να διέπουν το ποινικό δίκαιο, η ενοχή, η νομιμότητα, το ότι πρέπει να είναι κατανοητό, ε, το δίκαιο, η νομοθεσία πρέπει να είναι κατανοητή, δεν πρέπει να υπάρχει αμφισημία στη νομοθετική διάταξη και ούτε πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ. Και τελευταία αρχή αλλά βέβαια ίσως οι καθηγητές να αναφέρουν και άλλα στοιχεία, έχουμε και την ε, αρχή της ε, συνοχής. Γενικά στην ε, βιβλιογραφία λέγεται ότι η συνοχή για το ποινικό δικαίωμα είναι ουσιαστικό στοιχείο. Είναι το ίδιο που ανέφερα και πριν, ότι οι ποινέ θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένε μεταξύ του. Δηλαδή δεν μπορείτε να έχετε μια πολύ ψηλή ποινή για ένα δίκημα χωρίς να δείτε τι σημαίνει αυτό για τα άλλα δικήματα, πλούς επειδή υπήρχε κατακραυγή και πρέπει φυσικά να δούμε πώς νομοθετούμε σε αυτόν τον οίκο αλλά και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Νομίζω θα σταματήσω εδώ, γιατί ανυπομονώ να ακούσω τις παρεμβάσεις των ε, υπόλοιπων ομιλητών. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ε, αυτά τα γνωστά πρόσωπα εδώ σήμερα. Να σας πω ότι είχαμε και μια πολύ καλή συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών και Φυσικά σας ευχαριστώ για την συνεισφορά των ονομάτων. Διευκόλυνε τη ζωή του εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιάνγκ για την εισαγωγή αυτή στα βασικά θέματα. Οι αρχές ε, είναι η ε, επικουρικότητα, το ultima ratio και ποιοι είναι οι στόχοι, οπότε θεωρώ ότι καλό θα ήταν τώρα να ακούσουμε τον πρώτο εισηγητή μας, τον κύριο Χέρνς Νίλσεν, ε, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, ε, του <clears throat> Συμβουλίου του, Συμβουλ... του κολέγιου του Μπρούζ από το 1996. Ευχαριστώ. Εδώ θα σας μιλήσω σαν καθηγητής. Έτσι θα απευθυνθώ σε αυτή την επιτροπή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και ιδιαιτέρως να βλέπω ο, τόσους πολλούς πολύ ε, γνωστούς Ευρωπαίους στον τομέα αυτό. Βέβαια έχω λιγότερο από 20 λεφτά και είναι δύσκολο να ε, παρουσιάσω και την εξέλιξη του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιρροή της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά θα το προσπαθήσω. Όταν ήμουν στο στρατό, ο <clears throat> λοχίας μου είπε ε, μπορεί να σου φαίνεται εύκολα τα πράγματα, αλλά όταν θα στα εξηγήσω θα καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει με την εξέλιξη του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε ε, τόσα άτομα τα οποία υπησέρχονται από το 1900. Ε, 57 έχουμε τις εξελίξεις του Σένιεν, έχουμε ε, σε ε, κάποιο επίποδο την εξέλιξη στην νοτιοανατολική Ευρώπη και ε, τα Ηνωμένα Έθνη και στα πλαίσια αυτά είχα συναντηθεί <clears throat> γιατί αυτό συζητούσαμε τότε ε, με ορισμένους από εσά και βλέπουμε πως όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη. Από τις αρχές του Νοεμβρίου 1993, δηλαδή πριν από λιγότερο από 20 χρόνια, έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε το θέμα του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έγινε για πρώτη φορά στη συνθήκη ε, της, ε, του Μαστρίχτ ήταν μια διακυβερνητική συνεργασία και κάποια στιγμή κοίταξα τις πρώτες 100 αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί εκ των οποίων ε, ε, ε οι περισσότερες, ε, οι 99 δηλαδή, ήταν μη δεσμευτικές και μόνο οι εκατοστή ήταν δεσμευτικοί. Οπότε κατά την ε, πρώτη επανάσταση με τη συνθήκη της, ε, του Άμστερνταμ όταν αρχίσαμε να σοβαρευόμαστε στον τομέα αυτό την 1η Μαΐου 1999 ε, δηλαδή λίγο παραπάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει έκτοτε και δεν ε, επηρέασαν όλα αυτά τα θέματα άμεσα τις εξελίξεις και ε, ε, απλώς συμπεριελήφθησαν στις συνθήκες το Eurojust και το δικαστικό δίκτυο <clears throat> και αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε επίσης σήμερα. Ε, έκτοτε είχαμε το Τάμπερε, τη Χάγη, την πρόοδο της Στοκόλμης, την ε, στρατηγική ε, της Στοκόλμης. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα και το Συμβούλιο σε, ορισμένα, σε ορισμένες περιόδους παρουσίαζε πολλά προγράμματα δράσης αλλά όχι τόσο πολύ δράση και ε, οι περισσότερες εξελίξεις ε, ε, υλοποιόντουσαν στα ακράτη μελη εκ των οποίων ορισμένα ήταν υπέρ ενός κράτους έθνους, εθνικού κράτους και βάσιζαν το ποινικό δίκαιο εις την κυριαρχία και αν εξετάσετε την κυριαρχία μπορείτε να δείτε τις, την γνωμοδότηση για τη συνθήκη της Λισαβόνας του συνταγματικού δικαστηρίου Δικαστηρίου της Γερμανίας όπου βλέπετε ε, πώς, ε, ε, ότι αναφέρεται 23 φορές το θέμα του που μας απασχολεί. Και επίσης βλέπουμε ότι υπήρξε προσπάθεια να γίνει κάποια ενοποίηση και υπήρχαν πολλά κράτη τα οποία συζήτησαν τον, τη δικαστική συνεργασία και ε, δημιουργήθηκε το Corpus Juris, το πρώτο ποινικό ευρωπαϊκό δικαστήριο και το πρώτος ευρωπαϊκός ποινικό κώδικας. Και όλα αυτά ε, συνοψίστηκαν στο συμβιβασμό του Άμστερνταμ για να δημιουργηθεί ο χώρος ε, ελευθερίας και δικαιοσύνης ε, και ε, τώρα έχουμε ένα νέο μήνυμα, δηλαδή να μην υπάρχει πλέον διμερή συνεργασία μεταξύ κρατών ε, μελών. Δεν πρέπει να καταργήσουμε μόνο τα σύνορα για τους εγκληματίες αλλά και για την ποινική δικαιοσύνη και να υπάρχει πλήρης αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ε, φτάσαμε στο θέμα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο και ε, υπήρχε το ε, διπλό δικαίωμα πρωτοβουλίας από το Άμστερνταμ και το Συμβούλιο αργούσε πολύ να λάβει αποφάσεις και πολλές φορές καταλήγαμε στον κατώτατο κοινό παρανομαστή. Οπότε ουσιαστικά ε, περιοριστήκαμε σε τέσσερις ε, τομείς όπου η συνθήκη της, ε, του Άμστερνταμ και μετά του Τάμπερε συνόψισαν ε, τα διάφορα θέματα, την κατάρτιση οργανισμών όπως το Eurojust και η Europol και ε, ορισμένα δίκτυα τα οποία λειτουργούν σαν το Ευρωπαϊκό ο δικαστικό δίκτυο και ε, το δικαστήριο για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, και υπάρχει μία διασυνοριακή συνεργασία. Αλλά αν δείτε ακριβώς τι έγινε στην περίοδο του Άμστερνταμ ε, βλέπετε ότι καταρτήσαμε ένα εντυπωσιακό πλαίσιο με 35 αποφάσεις πλαίσιο που έχουν υιοθετηθεί και οδηγίες μαζί ε, εκ των οποίων 16 αναφέρονται στη συνεργασία, 12 ε, για την ε, αμοιβαία αναγνώριση, ορισμένες για την ουσία του ποινικού δικαίου και 5 οδηγίες. Δηλαδή Πρόκειται για ουσιαστική προσφορά από πλευράς ποσοτικής. Υπάρχουν επίσης 17 αποφάσεις για την κατάρτιση της Eurojust και της ε, ε, συνεργασίας για την εφαρμογή του νόμου ε, και δεν θέλω εδώ να επεκταθώ στις συστάσεις και στα ψηφίσματα. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό πλαίσιο νομοθετικό το το οποίο καταρτίστηκε κατά την περίοδο της συνθήκης του Άμστερνταμ και είναι κάτι το οποίο ε, ε, περιλαμβάνει 7 ή 8 δεσμευτικές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν τότε αλλά είχαμε ένα διτό πρόβλημα την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και τον έλεγχο της εφαρμογής. Όταν λοιπόν διαπραγματευτήκαμε τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ανέλαβε ορισμένα καθήκοντα γιατί προηγουμένως ε, στο Μάστριχτ, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστριχτ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε καν το δικαίωμα πρωτοβουλίες. Και τότε έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις. Το μόνο, τότε το Κοινοβούλιο είχε μόνο συμβουλευτικό ρόλο στα πλαίσια ε, του ε, δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, υπήρχαν δεσμευτικές αποφάσεις χωρίς όμως άμεση επίπτωση αλλά έμεση επίπτωση τη δυνατότητα δηλαδή του ποινικού δικαίου να υποχρεώσει τις εθνικές νομοθεσίες να συμμορφωθούν προς τις αποφάσεις αυτές που ήταν δεσμευτικές και ε, στο νομίζω ότι ε, στη συνέχεια προχωρήσαμε καλύτερα και συμμετείχαν 18 κράτη-μέλη. Μετά ε, περιελήφθη ο τρίτος πυλώνας, τον πρώτο πυλώνα, αλλά ακόμη σήμερα αμφισβητούμε εάν ε, υπάρχει μεγάλη επιρροή του τρίτου πυλώνα, διότι είναι μία ανάμνηση του τρίτου πυλώνα στον πρώτο πυλώνα. Έχουμε δηλαδή ορισμένους συσχετισμούς που αναφέρονται ή στο ποινικό δίκαιο και ε, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα κοινή και σημεριζόμενης ε, αρμοδιότητος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ακόμη δεν έχουμε εξετάσει όλες τις νομικές επιπτώσεις και επιπλέον ε, υπάρχουν οδηγίες και κανονισμοί στον τομέα αυτό δηλαδή έχουμε δυνατότητα δυνατότητα να καταρτήσουμε κανονισμούς δεν το έχουμε πράξει μέχρι στιγμής, θα γίνει στο μέλλον. Κανείς δεν σκέφτηκε λοιπόν τι σημαίνει να υπάρχει μία οδηγία ή στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Δεν μπορεί να έχει άμεσο ε, άμεσες επιπτώσεις εάν μιλάμε για ουσιαστικό δίκαιο και ε, σχετικά με την συνεργασία προς τα, ε, προς τα θύματα που μπορεί να έχουν άμεση επίπτωση στην εφαρμογή. Ιδίω όταν μιλάμε για την υυξημένη συνεργασία σε ορισμένα θέματα όμως δεν έχω δει ακόμη, ακόμη κάποιο αποτέλεσμα και ίσως κάποιος το εξετάσει και συντάξει κάποιο κείμενο μετά από την πρότασή μου σήμερα. Εξ όλων ε, αυτών όμως των δυνατοτήτων ε, υπάρχουν όλο και λιγότερες πρωτοβουλίες. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ενισχυθεί μετά από πέντε χρόνια, δηλαδή από την 1η ε, Δεκεμβρίου 2014 το Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν πλήρεις εξουσίες όπως προηγουμένως στον πρώτο πληλώνα για να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και να διατηρήσουν το νομικό πλαίσιο αλλά συγχρόνως να εφαρμόζουν τις αποφάσεις αυτές. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνη θα έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόζουν ήδη αυτές τις αποφάσεις. Όσον αφορά τη συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην μπορεί πλέον κανείς να αμφισβητήσει τη δημοκρατική νομιμότητα αυτών των αποφάσεων είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε από κοινού ε, το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε και ε, τη δυνατότητα του opt-out, μάλλον opt-in, δηλαδή ορισμένα κράτη μπορούν να αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν σε ορισμένες αποφάσεις. Η Δανία έχει μείνει απ' έξω αυτή την εποχή και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, ε, μπορώ να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό λέγεται ότι είναι δικό μου επινόημα αλλά το πρόγραμμα της Στοχόλμης εάν το εξετάσετε θα δείτε ότι του συμπεριφέρουμε σαν να είναι το μωρό μου μεν αλλά ε, πρόκειται για τις προσπάθειες της Σουηδικής Προεδρίας την οποία συμβούλευα εκείνη την εποχή είχα αυτή την τιμή. Και ε, σε σχέση με το παρελθόν προσπαθήσαμε να τονίσουμε περισσότερα τα θέματα της προστασίας ε, των ε, ατόμων, των στοιχείων, να μην εκτελούμε μόνο κατασταλτικές δραστηριότητες αλλά και πιο ήπιες δραστηριότητες που είναι προς όφελος των πολιτών. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα της Στοχόλμης, ήταν προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Αλλά υπάρχουν και πολλά κατασταλτικά στοιχεία και τονίσαμε ορισμένους τομείς προτεραιότητας και μπορούμε να δούμε ότι τώρα έχουμε προσυζήτηση πολλά θέματα τα οποία έχουν καθοριστεί από το πρόγραμμα της Στοκόλμης και θεωρούνται προτεραιότητες ε, ενίσχυση των ε, ατόμων, ε, κυβερνοέγκλημα και όλοι αυτοί οι τομείς τους οποίους έχουμε εξετάσει. Όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, η συνθήκη της Λισαβόνας λέγει ότι πρέπει να λαμβάνουμε δικαστικές αποφάσεις και να τις επεξεργαζόμαστε και αυτό δεν έχει ε, σύμφωνα με την, ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης τονιστεί τόσο πολύ όσο η αστυνομική συνεργασία. Εδώ μιλάμε για δικαστικές αποφάσεις οι οποίες σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον να καθοριστούν από τις αρχές οι οποίες θεωρούνται αυτούσιες τώρα πρέπει να επικυρωθούν οι αποφάσεις αυτές και να υπάρξει συνεργασία για την εκτέλεση και μιλάμε για διασυνοριακή διάσταση, όχι διασυνοριακές επιπτώσεις των αποφάσεων θα δείτε ότι ο όρος ε, διασυνοριακών ε, επιπτώσεων υπάρχει στο αστικό δίκαιο και στο ποινικό δίκαιο υπάρχει ένας ευρύτερος όρος ο οποίος εσκεμμένος έχει επιλεχθεί για να υπάρχει ευρύτερη συνεργασία από ό,τι στο αστικό δίκαιο. Δηλαδή υπάρχει μία, πολλές φορές μία διασυνοριακή διάσταση η οποία δεν συνεπάγεται ε, άμεσα άμεσα μία διασυνοριακή επίπτωση και προσφάτως έχω γράψει ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσα αγγλικά σε, ε, μία, σε ένα σουηδικό περιοδικό νομικό και μπορώ να σας το στείλω εφόσον είναι αγγλικά και λέγω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να λάβουν ορισμένες αποφάσεις γιατί ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε ε, μοιρασμένες αρμοδιότητες στα πλαίσια της ενώσεως και άπαξ και η Ένωση εξασκήσει τις αρμοδιότητές της δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του κράτους μέλους και νομίζω πλέον ότι οι άνθρωποι είναι θέμα της Ένωσης και ε, γι' αυτό παρόλο που θα αμφισβητηθεί σε 27 Υπουργεία Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάποια κάποια μέρα θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης της Ενώσεως. Και επιπλέον υπάρχουν ορισμένα αδικήματα τα οποία ποινικοποιούνται ε, λόγω της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όχι όμως λόγω αμελίας. Η αμέλεια για να θεωρηθεί ποινική θα πρέπει ε, να έχει άμεση επίπτωση στα κράτη-μέλη μέσω οδηγιών που θα έχουν άμεση εφαρμογή ε, και επιπτώσεις εάν δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά και ο συνάδελφος από την Πολωνική Προεδρία θα αναφερθεί στις ε, διατάξεις ε, ε, για, πιο πολύ ποινικό δίκαιο και έτσι δεν θέλω να προκαταλάβω τα δικά του τα λεγόμενα και απλώς να σας πω ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις διατάξεις ποινικού δικαίου. Έχουμε δηλαδή μεγάλη ευελιξία, πολλές δυνατότητες, αλλά όταν στη Σουηδική Προεδρία διαπραγματευθήκαμε το σημαντικό αυτό έγγραφο, είχαμε προβλέψει ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα, να υπάρξει κάποια συνεκτικότητα σε σχέση με ε, τις ε, ε, οδηγίες τις οποίες έχουμε υιοθετήσει και προφανώς θα χρειάζεται περισσότερη συνοχή στις σκέψεις και στις πράξεις μας. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ελπίζω ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν να υπάρξει και μεγαλύτερη συνεκτικότητα στο συνολικό τομέα. Και η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει νέες δυνατότητες όταν πρόκειται για αξιολογήσεις, για εκπαίδευση, ιδίω δικαστικού προσωπικού και είναι λυπηρό ότι υπάρχει τώρα μία αστυνομική ακαδημία σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να υπάρχει μία ευρωπαϊκή δικαστική ακαδημία ακαδημία η οποία θα έπρεπε να υπάρξει. Ε, έχω μεγάλες προσδοκίες για τις οικονομικές προοπτικές τις οποίες θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε 800 εκατομμύρια τα οποία διατίθενται στη δικαιοσύνη ενώ το 96 όταν ξεκίνησα μιλούσαμε για ένα πρόγραμμα για όλο το χώρο της δικαιοσύνης ύψους 2 εκατομμυρίων. αλλά βλέπετε ότι υπήρξε σημαντικότατη εξέλιξη. Ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο, στη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια και έχουμε και τον Ευρωπαίο Δημόσιο Εισαγγελέα, ο οποίος δεν ε, είναι, δεν είναι θέμα αν πρόκειται να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί, αλλά το ερώτημα είναι εάν θα υλοποιηθεί πριν ή μετά τη δικιά μου συνταξιοδότηση. Θα δούμε. Ας συζητήσουμε περισσότερο τι ε, συζητείτε τώρα. Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, παραδείγματο χάρη, θα υιοθετηθεί πολύ σύντομα. Έχουμε ε, ένα ένταλμα ερευνών ευρωπαϊκό, το οποίο ελπίζω ότι θα αντιμετωπίσει αντιμετωπιστεί θετικά στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα για να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Θα αρχίσουμε συζητήσεις με το Κοινοβούλιο για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που θα αρχίσουν στην επόμενη χρονιά. Έχουμε το θέμα των PNR, δηλαδή των προσωπικών δεδομένων που συζητείται και η ανταλλαγή τους. Η αμέλεια είναι σημαντικό θέμα. Έχουμε τα δικαιώματα των θυμάτων και ελπίζω ότι επίσης την επόμενη εβδομάδα θα διατυπωθεί μια κοινή προσέγγιση βάσει της πρωτοβουλίας της Πολωνικής Προεδρίας. Τα ουσιαστικά δικαιώματα για πληροφόρηση των υπόπτων οι οποίοι κατηγορούνται σε ποινικέ διαδικασίες και έχουμε αρχίσει να μιλάμε ε, και για εκμετάλλευση του χώρου και εκμετάλλευση ε, ε, διαφόρων πληροφοριών που θα έπρεπε να είναι εμπιστευτικές. Επίσης όσον αφορά τις κατασχέσεις, τις, τα προσωπικά στοιχεία, τα ευάλωτα άτομα, την το, διακίνηση να την προστασία δεδομένων, την αποζημίωση των θυμάτων, την ε, ε, κατάσχεση των οικονομικών πόρων ορισμένων τρομοκρατών, τα αναζητούμενα παιδιά, ε, η πολίτες τρίτων χωρών. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, τα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Βλέπετε ότι έχουμε μέχρι 20 σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που ε, ελπίζουμε να εξελιχθούν εντός των επομένων 18 μηνών. Ελπίζω λοιπόν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα ανοίξει νέες προοπτικές για μας και ότι ε, θα μπορέσουμε να έχουμε μία συνεργασία όχι μόνο πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν θα υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα και ότι ε, το Συμβούλιο και ε, το Κοινοβούλιο θα συνεργάζονται βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το ποινικό δίκαιο. Ευχαριστώ τον καθηγητή Νίλσεν. Σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε μια πραγματική εικόνα από τα μέσα όλης αυτής ε, της επανάστασης και ε, από ό,τι φαίνεται η καταπολέμηση του εγκλήματος έχει καταστεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Αναφερθήκατε σε θέματα όπως εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση των γυναικών, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, παραχάραξη, όπλα, ναρκωτικά, διαφθορά, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και καταπολέμηση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι μας ε, δώσατε επαρκή όθηση για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα, αλλά να ορίσω τον κύριο Αλ Γουίλιαμς, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, της ε, Eurojust Χαιρόμαστε που περιβρίσκεστε και πάλι εδώ. Πολλές φορές ε, έχετε παρευρεθεί στις ακροάσεις που οργανώνει η δική μας επιτροπή και πολύ χρήσιμη παρουσία σας σήμερα. Έτσι λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο σημείο που θα τον αναπτύξει ο κύριος Αντρέ Κλίπ, ο οποίος είναι καθηγητής ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και διακρατικού ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα τον κύριο Ντεγιόγκ για την πρόσκλησή του. Για μένα είναι μεγάλη τιμή η παρουσία μου ενώπιόν σας για να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω το ιστορικό της συνθήκης της Μαστρίχτης. Τα έχουν πει άλλοι, ο προηγούμενος δηλαδή. Μου ζήτησαν να πω μερικά λόγια για τις συνθήκες υπό τις οποίες το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο απαιτείται, είναι απαραίτητο. Ουσιαστικό μάλιστα ποινικό δίκαιο. Και εδώ τίθεται το συμπληρωματικό ερώτημα Ποια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται για να ισχύσει ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Τι κριτήρια ισχύουν όταν υπάρχει απόφαση δίωξης ευρωπαϊκά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Λόγω της αυξανόμενης σημασίας που έχει το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και θα έχει στο μέλλον, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτό το λέω γιατί μερικοί μπορεί να υποστηρίζουν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ρόλο και άλλοι να είναι αντίθετοι. Δεν πιστεύω όμως ότι οι εγκληματίες, κανείς δεν πιστεύει ότι οι εγκληματίες θα περιοριστούν στα εθνικά σύνορα και όρια. Γιατί μερικά εγκλήματα έχουν από τη φύση τους διαμεθοριακό χαρακτήρα. Για τις διώξεις τα κριτήρια τρία είναι, τρεις είναι οι συνθήκες. Πρώτον, να υπάρχει αποδεδειγμένη ζημία ή βλάβη. Συχνά στο ποινικό δίκαιο χρησιμοποιούμε γερμανική ορολογία Rechtsgut. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει αποδεδειγμένη με τον νόμο παρανομία και αδίκημα και ζημία. Δεύτερον, το ποινικό δίκαιο είναι το καταλληλότερο μέσο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το έγκλημα. Και τρίτον, αυτό που θα με απασχολήσει περισσότερο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εφαρμοστεί αντί της εθνικής, αυτό έχει προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για το Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, να διατυπώσει ρητά αυτά τα κριτήρια, έτσι ώστε να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία μερικός και ανεπαρκός όπως έγινε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτά που έχει προβλέψει το Συμβούλιο είναι χρήσιμα. Για το πρώτο κριτήριο, να αποδεδειγμένη ζημία ή βλάβη δηλαδή, δεν, αυτό δεν σηκώνει πολλή συζήτηση. Μερικές φορές βέβαια όταν πρόκειται για την παιδική πορνογραφία λέγεται ότι στόχος είναι η δίωξη να καταπολεμήσει ακριβώς τη διάδοση του φαινομένου. Άρα αρκεί εδώ να πούμε ότι δεν συζητιέται το κατά πόσον είναι βλαβερή η δραστηριότητα αυτή. Θα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο αν η εφαρμογή ενωσιακού ποινικού δικαίου είναι κατά το καταλληλότερο μέσον. Εδώ πρέπει να δούμε αν υπάρχει κανένα άλλο μέσο δίωξης που να μην αρκεί. Άρα χρειάζονται περισσότερα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το εθνικό ποινικό δίκαιο δεν μπορεί να καταπολεμηθεί δεν μπορεί να καταπολεμήσει επαρκώς μερικά εγκλήματα χωρίς ενωσιακή παρέμβαση. Υπάρχουν όμως πολύ λίγα στοιχεία για τέτοιου είδους δικαιοδοσίες και υπάρχουν και μερικές παγίδες που πρέπει να τις προσέξει ο νομοθέτης. Θα μπορούσαμε να πούμε από το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αδικήματα και εγκλήματα ότι φταίει το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο καθεαυτό. Γιατί βλέπουμε βιασμούς, κλοπές στα κράτη-μέλη που μπορούν να αντιμετωπιστούν εθνικά. εφόσον πάντα θα υπάρχει έγκλημα. Το γεγονός ότι σημειώνονται αδικήματα και εγκλήματα δεν λέει καθε αυτό ότι το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο δεν αρκεί για την αντιμετώπιση τους. Ως καθηγητής αλλά και ως ε, δικαστής στο εφετείο έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές προβλήματα που δείχνουν ότι Υπάρχει πολλαπλή νομοθεσία για το ίδιο θέμα όπως για το δουλεμπόριο και την εμπορία ανθρωπίνων όντων. Γιατί η νομοθεσία έχει αλλάξει και τροποποιηθεί τόσο πολλές φορές που καμιά φορά υπάρχουν επικαλύψεις. Συχνά είναι καλύτερο να αλλάξει εκβάθρον η νομοθεσία αντί να μπαλώνεται συνεχώς με πρόσθετη νομοθεσία. Έχουν γίνει, χρειάζονται εδώ σοβαρές αξιολογήσεις που να δείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικού ποινικού δικαίου σε, για πολλά θέματα που συζητιούνται όπως ε, και αυτό δείχνει μάλλον μέχρι τώρα από τις συζητήσεις φαίνεται ότι δεν είναι πρόβλημα ουσιαστικού ποινικού δικαίου αλλά δυνατότητας δίωξης και εφαρμογής του τελευταία αξιολόγηση της Κομισιόν αναφέρει ότι η σημασία δίνεται κυρίως στο κατά πόσον είναι βλαβερό το έγκλημα μάλλον παρά κατά πόσον είναι ανεπαρκές το ποινικό δίκαιο. Ας πούμε πόσα χρειάζεται να χάσει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος για να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Αυτό δεν λέει βέβαια ότι είναι ανεπαρκές το δίκαιο. Στις μελλοντικέ αξιολογήσεις νομίζω πρέπει να αναφέρουμε και ποιος είναι ο στόχος της νομοθεσίας. Πολλές φορές εμείς οι ακαδημαϊκοί έχουμε την εντύπωση ότι ο στόχος είναι να απαγορευτεί η δυνατότητα να σημειωθούν καν αδικήματα. Πρόληψη δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό στόχος. Θα σας πω μερικά λόγια τώρα για το τρίτο κριτήριο που νομίζω είναι το σημαντικότερο γιατί τα πρώτα δύο είναι, εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη ήδη ως γενικός κανόνας. Το τρίτο όμως κριτήριο είναι κατά πόσον είναι ωφέλιμο να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εδώ η βάση είναι η αρχή της επικουρικότητας, το πιο σημαντικό κριτήριο για τη συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι ωφέλιμο να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε περιπτώσεις όπου υπάρχει καθαρό ευρωπαϊκό καθαρός ευρωπαϊκός χαρακτήρας του ίδιου του εγκλήματος και άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε εθνικό απλώς ποινικό δίκαιο όπως το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος εφόσον δηλαδή το έγκλημα βλάπτει την ίδια την Ένωση στο σύνολό της. Η σταθερότητα του ενωσιακού νομισματικού συστήματος ή η προστασία του ευρώ είναι θέμα τέτοιου καθαρά πανενωσιακού χαρακτήρος. Η φύση δηλαδή του εγκλήματος, ιδίως του διεθνικού εγκλήματος, απαιτεί ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του. Η παιδική πορνογραφία θα μπορούσε να είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ τέτοιου διεθνικού εγκλήματος. Στην τελευταία της ανακοίνωση σχετικός η Κομισιόν αναρωτήθηκε για το κατά πόσον υπάρχει προστιθέμενη αξία στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και ανέφερε τέσσερις λόγους. Πρώτον, κοινό ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών γιατί δεν είναι πάντοτε πεπισμένοι ότι είναι ωφέλιμο να υπάρξει ευρωπαϊκή ενωσιακή ποινική νομοθεσία αφού υπάρχει η εθνική. Δεν εμποδίζει αυτό την ελευθερία κινήσεων των εθνικών διοκτικών αρχών. Δεύτερον, το ενωσιακό ποινικό δίκαιο μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα κρύβονται οι εγκληματίες πίσω από παράθυρα της εθνικής νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να δείχνουν ότι οι διαφορές στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο λαμβάνονται υπόψη από τους εγκληματίες. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι προσπαθούν να αποφύγουν τη σύλληψη. Αυτό είναι φανερό. Τρίτον, η αμοιβαία αναγνώριση του εγκληματικού χαρακτήρα. Δεν είναι πιστικό να δούμε πώς διαφέρει το ποινικό δίκαιο μεταξύ χωρών μελών, ενώ παράλληλα υπάρχει ενωσιακό ένταλμα σύλληψης. Και τέταρτον και τελευταίον, πιο πιστικό κριτήριο, ένα ενωσιακό ποινικό δίκαιο θα είχε χαρακτήρα πρόληψης κυρίως και αποτροπής. Αυτό είναι φανερά ωφέλιμο διότι είναι φανερό ότι ωφελεί την ζωή της ίδιας της ολόκληρης της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίφημη απόφαση του για την ακύρωση δύο άλλων αποφάσεων για την μόλυνση ορισμένων πηγών δείχνει ότι όποτε η επιβολή ενωσιακής κύρωσης θα καταλήξει σε προφανή αποτροπή ή πρόληψη μελλοντικών εγκλημάτων είναι φανερό ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Θα αναφέρω τώρα ορισμένες παγίδες που <clears throat> μπορεί να αντιμετωπίσουν οι νομοθέτες ως προς την ποινική νομοθεσία στην Ένωση. Το ερώτημα είναι το πρόβλημα οφείλεται σε ελλείψεις του εθνικού ποινικού δικαίου ή όχι. Παραδείγματος χάρη το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και οι στρεβλώσεις των αγορών. Πολλές φορές έχουν υπάρξει αθωώσεις και άλλες φορές δεν έγινε καν δίωξη γιατί ε, υπάρχουν ελλείψεις στο εθνικό ποινικό δίκαιο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα δεν έγκυται στο εθνικό ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Σε περιπτώσεις ενωσιακών, πανουσιακού χαρακτήρα απατών είναι φανερό ότι χρειάζεται μια πιο ενωσιακή νομοθεσία ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πολιτικός χαρακτήρας του αδικήματος μπορεί το εθνικό ουσιαστικό ποινικό δίκαιο να μην βοηθάει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα η οδηγία 2009-52 για τις κυρώσεις ε, των εργοδοτών σε περίπτωση αδικήματος από εργαζόμενο χωρίς καν να έχει καταδικαστεί από εθνικό δικαστήριο. Σε περίπτωση ας πούμε δουλεμπορίας. Εδώ καμία διοκτική αρχή δεν θα άρχιζε δίωξη με τέτοια βάση γιατί δεν υπάρχει σαφής ορισμός του ποινικού χαρακτήρα αυτού του αδικήματος. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας νέος ορισμός που να το επιτρέπει. Πολλές διατάξεις σε οδηγίες και σε αποφάσεις πλαίσια θεωρούν ότι ο ενωσιακός νομοθέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει δίωξη αυτεπαγγέλτος, ενώ δεν ισχύει αυτό. Γιατί πολλές λεπτομέρειες σε περιπτώσεις συμμετοχής και προετοιμασίας εγκλημάτων δεν μπορούν και δεν πρέπει να προβλέπονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ας καταλήξω τώρα με τις περιπτώσεις όπου ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο θα έπρεπε να τύχει νομοθεσίας. Θέματα δηλαδή που μπορούν να, όπου μπορεί να εφαρμοστεί ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Τα κριτήρια που ανέφερα να υπάρχει πραγματική βλάβη και ζημία, να μην υπάρχει επαρκής απάντηση από το εθνικό ποινικό δίκαιο και να έχει προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν ισχύουν αυτά τα κριτήρια, τότε θα ήταν χρήσιμο και απαραίτητο κιόλα να υπάρξει νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη έρευνα. Άρα χρειάζεται περισσότερη εγκληματολογική έρευνα για να υποστηρίξουν και τα κράτη-μέλη την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Πράγμα που τελικά θα σέβεται και την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της ultima ratio. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία καθηγητά. Μας παρουσιάσετε μια πολύ πιστική παρουσίαση και τα καταφέρατε και μέσα σε 15 λεπτά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν τώρα Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή Αγκάνια το Μαρτίν, που είναι καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Καστιγιαλαμάντσα, Μάντσα, στη Μαδρίτη. Ο καθηγητής θα μας παρουσιάσει το οικονομικό ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο, αλλά το Πανεπιστήμιο Καστιγιαλαμάντσα δεν είναι στη Μαδρίτη, είναι στο Τολέδο. Τι να σας πω, εγώ το ξέρω, αλλά το έγραφε εδώ και όταν το διάβασα αναγνώρισα το λάθος. Γιατί η Καστίγια Μάλτσα δεν είναι στη Μαδρίτη, φυσικά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που οργανώνετε ε, αυτό το βήμα διαλόγου μεταξύ πανεπιστημίου και νομοθετών, επιστημίων και νομοθετών. Ε, νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα για μια συνεκτική νομοθεσία. Εγώ θα διαιρέσω την παρουσίασή μου σε τρία μέρη. Καταρχήν, θα κάνω μία σύντομη παρουσίαση της απόψης μου για το πώς ε, ε, πρέπει να ρυθμίζουμε κυρίως το οικονομικό έγκλημα. Κατόπιν θα δώσω κάποια παραδείγματα γιατί δεν προχωρήσαμε έτσι όπως ε, αναφέρουν οι συνθήκες και στο τρίτο μέρος ε, θα ήθελα να προβληματιστούμε για το εξής. Ποια είναι η αξιολόγηση της νομοθεσίας. Από τη δική μου οπτική η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι σαφής. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό έγκλημα, οι συνθήκες επιτρέπουν επιτρέπουν και μας υποχρεώνουν ε, να έχουμε ε, μία λογική ποινική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, κάποια βασικά στοιχεία για μια εξορλιστική ποινική πολιτική. Καταρχήν να υπάρχει αρμοδιότητα παρέμβαση σε οποιοδήποτε πρόβλημα που ανακύπτει σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπου έχουμε διασυνοριακό έγκλημα. Το κατακαιρματισμένο ποινικό δίκαιο είναι ένα άλλο λόγο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λόγο να έχουμε κατακαιρματισμένη πολιτική. Κατά την άποψή μου, το οικονομικό ποινικό δικαίο είναι ο τομέα όπου απριόρι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες ε, για να δημιουργήσει μια κοινή ποινική πολιτική. Οι συνθήκε επιτρέπουν ευρεία παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των οικονομικών εγκλημάτων. Έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα παρέμβασης. Ε, καταρχήν, το μοντέλο της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων αυτό είναι το πιο ισχυρό μοντέλο. Ευρωπαίος ε, δημόσιος κατήγορος, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω εναρμόνιση, υπάρχει ε, δυναμία να χρησιμοποιηθεί το emergency break ε, και ε, για τους λόγους αυτούς θα ήταν αδύνατο να δημιουργήσουμε οικονομικό ποινικό δίκαιο, ομοσπονδιακά δηλαδή εγκλήματα. Έχουμε και το άρθρο 83, το οποίο θα μπορούσε να διαιρεθεί σε τρία μέρη. Το 83.1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ του οικονομικού εγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος. Και σε ορισμένου ε, τομείς ε, είναι συχνό. Παίρνουμε το σχάρι όταν έχουμε παράνομη διακίνηση αποβλήτων. Όμως έχουμε και το άρθρο 83.2 το οποίο επιτρέπει ισχυρότερη παρέμβαση. Αυτό η προπόθεση προποθέτει ότι τα, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν ε, τις ε, κατάλληλες κυρώσεις για οποιαδήποτε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κάτι τέτοιο ισχύει σε άλλου τομεί, παραδείγματο χάρη στην τρομοκρατία και στην παιδική πορνογραφία. Οι οδηγίε καθορίζουν ποιε συμπεριφορέ απαγορεύονται και ποιε κυρώσει επιβάλλονται. Όμως, στην περίπτωση του 23.2, 2, όπως και στην περίπτωση της οδηγίας που αφορά την ε, ευθύνη σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ε, τέτοιες ε, συμπεριφορές μέσα στον κανονισμό και εδώ η εναρμόνιση αφορά κυρίως τις ποινές, τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Και τρίτον, αν χρειάζεται παρέμβαση στον τομέα των ε, οικονομικών εγκλημάτων. Ε, οι διατάξεις που προβλέπονται στο 83.1, στο δεύτερο τμήμα, μπορούν παντού να χρησιμοποιηθούν. Το δεύτερο στοιχείο της ε, λογικής της ευρωπαϊκής ποινικής πολιτικής είναι να υπάρχει ίση κατανομή των αρμοδιοτήτων σε εθνικό και περιεθνικό επίπεδο και έχουμε τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Αν ε, μιλήσουμε σοβαρά για τις αρχές αυτές, ε, τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, παρέμβαση στον ε, τομέα του εθνικού ποινικού δικαίου. Αυτό δεν πρέπει φυσικά να οδεύει προς εναρμόνιση. Το άρθρο 83 αναφέρεται σε εναρμόνιση, όμως αν ληφθούν υπόψη αυτές οι αρχές ε, θα πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική στην εναρμόνιση προκειμένου να, βρεθούμε σε μια, να βρούμε μια κοινή προσέγγιση για τα κοινά προβλήματα. Θα πρέπει η εναρμόνιση να είναι το έσχατο μέσο, τη μαράσιο της παρέμβασης για την αντιμετώπιση ενός ε, προβλήματος ε, κοινής εγκληματικότητας. Όμως, η λύση δεν θα πρέπει να είναι είτε εναρμόνιση είτε τίποτα. Όπως ανέφερα πριν, το πρόβλημα δεν είναι ο ορισμός των συμπεριφορών που πρέπει να απαγορεύονται, αλλά να καθορίσουμε τη φύση των ε, ποινών που πρέπει να επιβάλλονται και πόσο αυστηρές ε, πρέπει να είναι. Εδώ έχουμε κάποιες ε, ιδέες, ε, ε, έχουμε το αρχές αναλογικότητας και τις υπηρεκορικότητες πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται σε τρία βήματα. Αποτελεσματική, οι αποτελεσματικέ κυρώσεις πρέπει πάντοτε να εξαρτώνται και από την αρχή από τα κράτη-μέλη. Υποχρεούνται να ε, θεσπίσουν αποτελεσματικές, ε, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Όπως ε, γνωρίζουμε φυσικά και έχουμε σοβαρή, πρέπει να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση και στην περίπτωση ε, που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, το κράτος μέλος που δεν συμμορφούται, ε, θα πρέπει να τιμωρηθεί μόνο όταν ε, υπάρχει σημαντικός λόγος για εναρμόνιση των κυρώσεων, τότε θα πρέπει να λαβεί χώρα αυτή η εναρμόνιση. Πάντως, όπως είπα, αυτός ο τρόπος πρέπει να είναι το έσχατο μέσο ultima Το τρίτο στοιχείο είναι να αποδείξουμε ότι οι επιδιωκόμενοι σταοχοί συνάδουν με τα ήδη φυστάμενα και με τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου. Αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί, θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι κυρώσει συνάδουν με ε, ότι υπάρχει σε άλλες οδηγίες, δηλαδή η κατάχρηση της αγοράς δεν μπορεί να τιμωρείται πιο αυστηρά από ό,τι μπορεί ανθρώπων και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνοχή και με την εθνική ποινική νομοθεσία από την παρέμβαση μου μέχρι τώρα θέλω να τονίσω ότι καταρχήν υπάρχουν δυνατότητες ε, παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, προβλέψει αποτελεσματικές αναλογικές και αποτρεπτικές ε, κυρώσεις για παραβιάσεις στο οικονομικό τομέα και ότι η εναρμόνιση είναι το έσχατο μέσο τη για την παρέμβαση. Όταν έχει αναλυθεί, αφόσον θα έχει αναλυθεί το ιδανικό πλαίσιο, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην πραγματικότητα για να δω πόσο καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα. Καταρχήν, πώς ε, οι αρχές αναλογικότητας και επικουρικότητας διαλογούνται ε, στον τομέα αυτό. Η απάντηση είναι πολύ άσχημα. Οι αρχές αυτές δεν αναφέρονται καν από την απόφαση πλαίσιο που αφορά την ε, διαφθορά στον τομέα του περιβάλλοντος και στον ιδιωτικό τομέα για την οδηγία για την κατάχρηση στην αγορά υπάρχει μία ρήτρα που αφορά το διασυνοριακό χαρακτήρα ε, του αδικήματος, αλλά είναι μία πρότυπη ε, διάταξη, μία πρότυπη ρήτρα. Ε, έχαμε και τις προσκευαστικές εργασίες βεβαίως και στην ε, περίπτωση του οικονομικού εγκλήματος το κύριο επιχείρημα είναι να αποφύγουμε τους περιορισμούς στην αγορά. Όμως το επιχείρημα αυτό το οποίο αναφέρεται γενικώ φέρνει δύο προβλήματα ε, έναντι της αιτιολόγησης της εναρμόνισης. Το πρώτο είναι εμπειρικό, όπως ήδη ανέφερα στα πλαίσια του οικονομικού ποινικού δικαίου Υπάρχει διαφορετικό επίπεδο αυστηρότητα των ποινών. Έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο κανονιστικού χαρακτήρα. Η χρήση τέτοιων επιχειρημάτων είναι επικίνδυνη γιατί ο τρόπος της διαχείρισής τους μπορεί να μας οδηγήσει σε περισσότερη ποινική νομοθεσία. Έτσι λοιπόν, αυτό που στρεβλώνει την αγορά ε, είναι οι χαμηλότερες ε, κυρώσεις. Αυτό θεωρείται βέβαια γι' αυτό το λόγο η εναρμόνιση τίνει να αυξάνει αυτές τις ποινές, αυτές τις κυρώσεις. Πρόσθετα, σύμφωνα με τα επιχείρηματα αυτά, αυτό που θα έπρεπε να κάνει η οδηγία είναι να προσπαθήσει να παρεμποδίσει το να υπάρχουν πιο αυστηρές κυρώσεις, ε, γιατί τότε θα μπαίναμε σε έναν κύκλο, φαύλο κύκλο και θα οδηγούμαστε σε περισσότερο ποινικό δίκαιο. Η ιδέα της εναρμόνισης των ελάχιστων προτύπων είναι ακριβώς αντίθετη σε αυτό. Και τα δύο προβλήματα μας οδηγούν σε κάτι που έχει φανεί εδώ και καιρό. Στην αναλογικό, η αποτελεσματικότητα των ποινών, αυτό είναι το πραγματικό αποτρεπτικό στοιχείο. Και αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω στην παρέμβασή μου. Οι διαφορές ε, στην αποτελεσματικότητα είναι αυτό που διαφοροποιεί τα διάφορα ποινικά συστήματα των κράτων μελών. Ένα παράδειγμα για την κατάχρηση στην αγορά. Η οδηγία αφήνει στα κράτη-μέλη ένα ευρύ διακριτικό πλαίσιο για την θέσπιση των κυρώσεων. Ως συνέπεια έχουμε διαφορετικές κυρώσεις. Ε, σε όλες τις χώρες ποινικοποιείται το insider trading και η ποινή μπορεί να είναι από ένα έτος στο Βέλγιο μέχρι στα 15 στην Ιταλία αν δούμε τις σχετικές συμπεριφορές σε ορισμένες χώρες υπάρχει ισχυρή παρουσία πενικού δικαίου και ε, διοικητικών κυρώσεων. Όμως, πέρα από τις διαφορές μεταξύ των κυρώσεων, αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον είναι η διαφορετική χρήση ε, αυτών ε, των ποινών στην ε, Ισπανία. Μετά από 12 χρόνια, μετά την πρώτη οδηγία για το insider trading, καμία ποινική κύρωση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη και μόνο μία φορά έχει υπάρξει μία περίπτωση για τέτοιο έγκλημα. Το ίδιο και θα γίνει και με την οδηγία για την κατάχρηση στην αγορά που πρόσφατα εισήχθη. Όμως το πρόβλημα δεν είναι το ποινικό δίκαιο, αλλά πώς ε, οι Ισπανικές αρχές παρακολούθησης ε, των χρηματαγορών ε, απαντούν σε αυτές τις συμπεριφορές. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η εναρμόνιση. Λοιπόν, να σχολιάσω και κάτι άλλο, πολύ σύντομα. Σίγουρα, ορισμένε φορέ το ποινικό δίκαιο προκαλεί στρεβλώσει στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, αυτέ τι στρεβλώσει δεν θα πρέπει να αποδίδονται στι ε, διαφορετικέ κυρώσει, αλλά στο τι διαφορετικό απαγορεύεται. Παραδείγματο χάρη, ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις στα νομικά πρόσωπα. Κάθε απόφαση, πλαίσιο, οδηγία και σύμβαση από το δεύτερο πρωτόκολλο του ε, το προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων θεσπίζει υπευθυνότητα, ευθύνη για τα νομικά πρόσωπα. Και τα κράτη-μέλη έχουν ε, ψηφίσει διάφορε κυρώσει σε κάποιε χώρε όπω η Ιταλία και η Γερμανία. Έχουμε και διοικητικέ κυρώσει. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι κυρώσει στην πράξη είναι τόσο αποτελεσματικές όπως και οι ποινικέ κυρώσει που εφαρμόζονται στην Γαλλία και στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα στον τομέα αυτό είναι, όπως θέλω να τονίσω, ότι υπάρχει έλλειψη ασφαλείας δικαίου. Οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν ε, να τους επιβληθεί κάποια κύρωση. Ενώ στην Ιταλία, στην Αυστρία, παραδείγματος χάρη, τα προγράμματα συμμόρφωσης ε, θεωρητικά ε, δεν χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες μάλλον σε εκείνες χώρες εφαρμόζονταν σε άλλες χώρες όπως τη Γαλλία δεν έχουν καμία αξία τα προγράμματα αυτά. Και αυτό είναι ακόμη πιο προβληματικό στις χώρες όπου τα προγράμματα συνόρφωσης ε, έχουν νομική σχετικότητα, ε, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία, υπάρχει απέτηση να δημιουργηθεί ένα όργανο εποπτείας χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό το τελευταίο παράδειγμα Μα δίνει κάποια διδάγματα σε σχέση με την εναρμόνιση. Καταρχήν, επικουρικότητα και αναλογικότητα, οι αρχέ αυτές δεν έχουν ε, πρακτική ισχύ ε, και δεν λαμβάνονται παρκώ υπόψη οι αρχές αυτές κατά την εκμόνιση των οδηγιών. Δεύτερον, ε, στην αγορά βλέπουμε κυρίως ότι υπάρχει διαφορετικά επίπεδα οικονομικού ποινικού δικαίου και ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό και όχι η ύπαρξη διαφορετικών κυρώσεων. Όπως ξέρετε δεν ε, είναι πανάκια κυρώσεις ε, για την αρρώστια αυτή. Τρίτον, η εναρμόνιση είναι απαραίτητη όταν υπάρχει έλλειψη ασφαλής δικαίου και όταν οι παράνομες συμπεριφορές δεν ποινικοποιούνται μάλλον και όταν οι συμπεριφορέ αυτέ είναι εντελώ διαφορετικέ και όχι όταν είναι διαφορετικές οι κυρώσει. Και θα συνεχίσω με το τελευταίο τμήμα τη παρεμβασή μου. Πώ ε, θα κάνουμε ό,τι αρμόζει στο μέλλον. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του ποινικού δικαίου. ορισμένε βασικέ ιδέε τώρα. Καταρχήν πρέπει το, να τα αξιολογήσουμε. Δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώνουμε αν ένα κράτος μέλος έχει με ακρίβεια εφαρμόσει την απόφαση πλαίσιο ή την οδηγία, όπως κάνει η Κομισιόν μέχρι τώρα. Η αξιολόγηση είναι κάτι πολύ πιο εκτεταμένο από αυτό. Δηλαδή, δεν πρέπει να αξιολογηθεί μόνο το θέμα της εναρμόνισης του νομικού δικαίου, αλλά οποιοδήποτε σχετικό τομέα πέρα από τον οικονομικό πρέπει να αξιολογηθεί. Επίση, ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιβολή τη νομοθεσίας και τα συγκεκριμένα προβλήματα τη εφαρμογή του νόμου. Επίση, στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πόσο έχουν ε, επιτευχθεί οι βασικέ αρχέ και πόσο έχουν γίνει σεβαστέ οι αξίε του ποινικού δικαίου. Επίση, ποιο είναι επικεφαλή αυτή τη αξιολόγηση, Πρέπει να υπάρχει ε, ένας ανεξάρτητος αξιολογητής, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την αξιολόγηση των ποινικών πολιτικών. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα διάφορα παρατηρητήρια από μια κοινή μεθολογία. Αυτός ο οργανισμός αξιολόγησης θα πρέπει να σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ασκεί τις ελεκτικές του εξουσίες. Και το να έχουμε διαφορετικές ελληνικές πολιτικές δεν μας επεξηρετεί. Οι αρχές δεν έχουν καμία αξία χωρίς την αξιολόγηση και χωρίς ε, ο νομοθέτης να έχει το βάρος της απόδειξη και την υποχρέωση να αποδείξει ότι η απαγόρευση, η κυρώσεις και γνωρίσει είναι απαραίτητες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τώρα αρχίζουμε <clears throat> το χώρο για συζήτηση και παρακαλώ όποιο <clears throat> θέλει να παρέμβει ε, να σηκώνει το χέρι του. Προτείνω λοιπόν να συγκεντρώνουμε μία σειρά ερωτήσεων και μετά το <clears throat> Προεδρείο να απαντήσει και ε, πρέπει να σας πω ότι κινδυνεύουμε να ξεπεράσουμε τα όρια μας Εξού και θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσουμε τώρα με την ερώτηση της κυρίας Λάτφορντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση ήταν όντω πολύ ενδιαφέρουσα και ε, την βρήκα και ανησυχητική. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις σοβαρές ε, προειδοποιήσεις τις οποίες ε, μας απευθύνουν οι ακαδημαϊκοί και καθηγητές. Ο καθηγητής ε, Κλικ είναι ένας δικαστής ο πρόκειται όλοι για σημαντικές προσωπικότητες και βλέπουμε ε, ότι ενώ ε, είχαμε καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα τώρα ερχόμαστε εις μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα κατατήσει μία επιτροπή να συζητηθούν ορισμένα θέματα όπως και ε, το θέμα των αποτρεπτικών κυρώσεων, το θέμα της συμπεγνίας και της βοηθείας και νομίζω ότι όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό και είμαι μετριοπαθής. Ο καθηγητής Κλίπ μας είπε ότι δεν θα ήταν δυνατόν κάποιος δικαστής ε, να ε, καταδικάσει και ε, κάποιον βάση της οδηγίας για την απασχόληση. Οπότε, εάν κατάλαβα καλά, Σύμφωνα με ε, το θέμα της ε, ε, προκατάληψης που προβλέπεται στο Ολλανδικό δίκαιο και μπορεί να αμφισβητηθεί σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τότε ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να ποινικοποιήσει την αμέλεια και ε, εδώ και πολύ καιρό νόμιζα ότι καλύπτουμε με τους εμπειρογνώμονες διάφορα θέματα ασχέτως των ε, επιπτώσεων που θα υπάρχουν εις ε, τις δικαστικές αποφάσεις δηλαδή πώς θα καθορίσουμε την ελάχιστη ή ανώτατη ποινή σε μία οδηγία. Αισθάνομαι λοιπόν και ταπεινωμένη και ε, ανήσυχη διότι δύο χρόνια μετά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το οποίο ε, ζητούσε από την Προεδρία να συζητήσει το θέμα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εγώ τουλάχιστον ε, δεν γνωρίζω να έχει έρθει οποιοδήποτε και να πει στο Κοινοβούλιο ότι παιδιά αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει σοβαρή συζήτηση και ε, ο κύριος Γιόγκο για την ε, ακρόασή του δυστυχώς έχει οργανώσει μία πέμπτη πρωί όπου όλοι έχουν γυρίσει σπίτια τους αλλά είναι πλέον επίγον να εξετάσουμε και να σταθμίσουμε τη σημασία του ο ποινικού δικαίου εις ε, την Ευρώπη και να δούμε ε, τι μπορεί να είναι ενδεχομένω οι επιπτώσεις που θα συμπαρασύρουν αυτές οι κινήσεις για τα οικονομικά εγκλήματα όπου δεν υπά... έχει υπάρξει ποτέ ένα σύστημα κυρώσεων. Ας μην προχωράμε στα τυφλά και ε, όντως πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει ε, από το τεράστιο όγκο των πληροφοριών που μας δόθηκαν σήμερα είμαι πολύ ευγνώμων αλλά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για το νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάποιο άλλο σχόλιο, ερωτήσεις, θέματα, δεν βλέπω. Οπότε δίνω το λόγο εάν ε, κάποιος θέλει να σχολιάσει τα θέματα τα οποία έθεσε η κυρία Λάτφορντ, ο κύριος Νίλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ είμαι και πολύ ε, ταπεινωμένος και ανήσυχος διότι δουλεύω εδώ και 25 χρόνια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το ποινικό δίκαιο που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που έχει καταρτιστεί ε, και συγκροτηθεί από τα εθνικά συστήματα που βασίζονται στην εδαφική κυριαρχία και υπάρχουν πολλά εγκλήματα, ιδίως αυτά τα οποία εντοπίζονται ή στη συνθήκη όπου επίγεται να ε, συνέλθουμε και να σκεφτούμε πώς θα εξετάσουμε από κοινού και θα καθορίσουμε από κοινού τα θέματα αυτά εφόσον μιλάμε για διασυνοριακή εγκληματικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με διακίνηση ανθρώπων, με ε, παραποιήσεις, καταχρήσεις και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και βλέπουμε ότι η ε, παραποίηση και η ε, διαφθορά είναι τα πλέον σοβαρά θέματα που πραγματεύεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται τα, εδώ και δύο χρόνια να ε, εμπλακεί, χρειάστηκε εδώ και δύο χρόνια να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω υπάρξει και παραστεί σε πολύ τριμερείς ε, συζητήσεις για να Trying αναμορφώσουμε τις πρακτικές μας και να διορθώσουμε τις πρακτικές ορισμένων κρατών τα οποία ακολουθούν λάθος δρόμο. Νομίζω ότι η αναφορά στην ανάπτυξη των διατάξεων του συγχρόνου ποινικού δικαίου το έγγραφο του Συμβουλίου της 30 Νοεμβρίου 2009 τονίζει ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την νομοθετική διαδικασία σε αυτή τη διεργασία και να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί. Δηλαδή, εάν υπάρξει ένας ορισμός μίας αξιόπινης πράξεως, συμμετοχή, συνεργία, συγκάλυψη, ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και να μην συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις απλώς μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να συνεχίσει. Χαιρετίζω την έκθεση που έχει καταρτιστεί και αποτελεί μέρος της διαδικασίας ότι χρειάζεται να συζητήσουμε το θέμα περαιτέρω όσον αφορά τις ε, κυρώσεις. Η συνθήκη μπορεί να μας επιτρέψει ε, να έχουμε κατά προσέγγιση κυρώσεις, αλλά ουσιαστικά ε, δεν έχουμε πολλά μέχρι στιγμής. Είπατε πολύ σωστά θα πρέπει να έχουμε ελάχιστη ή ανώτατη κύρωση για την τρομοκρατία που να είναι 8 ετών σε άλλες χώρες χώρες είναι πολύ ψηλότερες. Οπότε αυτό δεν έχει μεγάλο νόημα και βλέπετε ότι έτσι δεν επηρεάζεται το κράτος μέλος ή ε, την ε, νομοθεσία σχετικά με την ε, απελευθέρωση, αποφυλάκηση υποαίρεση ή ε, υπό συγκεκριμένε συνθήκες. Άρα εάν ήμασταν όντως σοβαροί θα έπρεπε να έχουμε προβεί σε μια διαφορετική διαμόρφωση του θέματος με ε, ε, βάση άλλες ε, αποδείξεις από αυτές που χρησιμοποίησαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε αρκετέ πληροφορίες για την εφαρμογή της ποινική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ λίγε πληροφορίε για την πραγματική χρήση τη νομοθεσία αυτή στα κράτη-μέλη. Και επομένως ε, έχουμε κάποιες ενδείξεις για τις αιτίε. Οι αιτίε θα μπορούσαν να είναι η λεπτομερής φύση της νομοθεσίας. Έδωσα ένα παράδειγμα. Δεν σκοπεύω να πω ότι όλες οι απαγορεύσεις ε, στην οδηγία που ανέφερα είναι τέτοια φύσεως. Έδωσα ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα και ουσιαστικά θα συμβούλευε οποιοδήποτε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ακολουθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ μπορώ να αναφέρω τώρα την ε, νομοθεσία για την απάτη που εφαρμόζεται πολύ σωστά από τις κατοχώρες στο εθνικό δίκαιο και υπάρχουν κάποια στοιχεία που ε, ουσιαστικά φορούν ε, την πυκνοποίηση επιφορών που ε, ουσιαστικά δρούν ε, εις βάρος του προβληξμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως υπάρχουν κάποιες άλλες διατάξεις που δεν χρησιμοποιούνται. Πετείται παραδείγματος χάρη ότι θα μπορούσε να αποδεικτεί ότι υπήρξε ε, παραχάραξη πριν χάρη και κάποια χρήματα κατευθύνθηκαν προς τα κάπου όπου δεν θα έπρεπε και κάποιος ε, σκόπιμα είχε κέρδος, Εποφελήθηκε από αυτό. Αυτό αρκεί και αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μια τέτοια διάταξη για τη δίωξη εγκλημάτων απάτης. Όμως αυτό δεν βλέπετε να αναφέρεται στατιστικές. Έτσι λοιπόν το μήνυμά μου είναι να διατηρήσουμε απλή την νομοθεσία στο ποινικό δίκαιο και να είμαστε ε, ουσιαστικά επικεντρωμένοι στον πυρήνα, τι θέλουμε να προστατεύσουμε και να μην προσθέτουμε διάφορα στοιχεία. Όλα τα διάφορα στοιχεία θα πρέπει να αποδειχτούν, ε, θα πρέπει κάποιο να ασκήσει δείξη και θα πρέπει να παρουσιαστούν και αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν εγγύσεις ότι θα έχουμε επιτυχία έκβαση στην υπόθεση. Ευχαριστώ κύριε Σνέντο Μαρτίν. Νομίζω ότι ο ορισμός δεν είναι το ουσιαστικό της ενεργόνησης. Μπορούμε να ορίσουμε τι επιθυμούμε, αλλά στη συνέχεια, όπως συμβαίνει και στο εσωτερικό μας δίκαιο, υπάρχουν πάρα, πολλές διαφορετικές, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και υπάρχει απόκληση από τη θεωρία στην πράξη. Νομίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ δύσκολο καθήκον να έχει ακριβώς ε, τις ίδιες έννοιες που θα ισχύουν σε όλε τι χώρε. Δεν είναι αυτό το καθήκον τη εναρμόνισης από την άποψή μου. Μιλάμε ε, ουσιαστικά για ισοδύναμη προστασία των ένομων συμφερόντων. Αλλά αυτό αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας, όχι την ίδια την νομοθεσία. Η ιδέα της οδηγίας είναι ε, μία ιδέα που σχετίζεται με την αξιολόγηση. Το σημαντικό σε κάποια οδηγία δεν είναι το κείμενο της ίδιας της οδηγίας, αλλά είναι ο στόχος της οδηγίας. Με αυτό κατά νου πιστεύω ότι η αξιολόγηση είναι ένα από τα πλέον σημαντικά. Πριν να κάνουμε ένα βήμα παρατέρω στην εναρμόνιση, νομίζω ότι η εναρμόνιση δεν αποτελεί καλή λύση για τα προβλήματα που έχουμε στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Α, ωραία. Ευχαριστούμε. Τώρα έληξε ο πρώτος γύρος. Περνάμε στον δεύτερο που θα είναι σίγουρα το ίδιο ενδιαφέρον και με το πρώτο. Με τον πρώτο. Πώς θέλετε να σχολιάσετε τίποτε εκεί πίσω. Ναι, αλλά τότε σύντομα παρακαλώ, γιατί καθυστερούμε, καθυστερούμε. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Ναι, ευχαριστώ. Αν αυτό ταιριάζει καλύτερα στους άλλους γύρους, να το αναβάλω. Είμαι ο βοηθός της Ευρωβουλεύτριας Μονίκα Μακοβέη. Φαίνεται ότι σε πολλούς τομείς μπορεί να γίνει ωφελήμος παρέμβαση ενωσιακός αλλά πρέπει να γίνει προηγουμένως μια αξιολόγηση. Καλά το κατάλαβα. Μιλήσατε για αξιολόγηση εφαρμοστικής, δηλαδή πώς λειτουργούν τα ποινικά συστήματα στα κράτη-μέλη, τα δικαστικά συστήματα, κατά πόσον είναι αποτελεσματικά, διαφανή κλπ. Τι κριτήρια θα χρησιμοποιούσατε, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Η αξιολόγηση είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά αρκεί να έχουμε μία πιο λογική εγκληματολογική πολιτική, πολιτική δίωξη του εγκλήματος η μεθοδολογία για την αξιολόγηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Είναι απαραίτητη μεν, αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε απλώς ότι δεν υπάρχει συνδυασμένη, εκλογικευμένη δίωξη του εγκλήματος. Στην Ισπανία η νέα κυβέρνηση προτείνει μακροχρόνια κράτηση πριν ακόμη από τη δίκη. Αυτό είναι παραλογισμοί. Αν γίνει ο απολογισμός η αξιολόγηση τότε τέτοιου είδους προτάσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Νόημα, πώς να το πω. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Θα προεδρεύσει ο, η αντιπρόεδρος Κίνγκα Γκόντς. Ελάτε εδώ να προεδρεύσετε παρακαλώ. Και οι ομιλητές επίσης να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Um, Καλωσορίζω τους ομιλητάς του δευτέρου μέρους. Ε, συνεχίζεται η ακρόαση γιατί βιαζόμαστε. Τι να χρησιμοποιήσω, αυτό, α ναι. ε, Έχουμε εδώ λίγους αλλά καλούς ευρωβουλευτάς. Πρώτα απ' όλα ο καθηγητής Ράιμο Λάχτη που είναι καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη θα λάβει το λόγο πρώτος και μετά θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπου. Πάρε, πάρε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, όντως είναι για μένα μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε αυτήν την συνεδρίαση και θα χρησιμοποιήσω ορισμένα, ε, ορισμένες διαφάνειες αλλά θα προσπαθήσω να παρουσιάσω διάφορα θέματα τα οποία ίσως ε, δεν συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση. Νομίζω ότι τώρα δουλεύει το μεχάνημα. Λοιπόν, πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως είπε και ο καθηγητής Νίλσον, ίσχυαν άλλα πράγματα που δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Αυτή η διαφάνεια πάντως που βλέπουμε εμείς ανάποδα εδώ ε, αφορά τις επικρίσεις που ακούγονταν πριν ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνος. Οπότε και δινόταν πολύ μεγάλη σημασία στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των νομοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τη Σκανδιναβία ακούγονταν επικρίσεις γιατί και εγώ από σκανδιναβική χώρα είμαι και ξέρω ότι πολλές φορές ακούστηκαν και μέσα στην Ένωση τέτοιες επικρίσεις. Παραδείγματος χάρη το ρόλος ότι δεν ήταν ανεπαρκής η πρόληψη του εγκλήματος και κριτήρια όπως η νομιμότητα και η ανθρωπιά δεν αναλαμβάνονταν επαρκώς υπόψη. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών κυρώσεων ως μέσο μάλλον αποτροπής παρά κύρωσης. Αυτά ήταν οι κύριες επικρίσεις που ακούγονταν στην δυναβία. Τώρα όμως υπάρχουν νέες εξελίξεις και νέες δυνατότητες. Και αυτό είναι πολύ θετικό για την εξέλιξη της ποινική πολιτικής, της εγκληματολογικής πολιτικής της Ένωσης. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει τώρα σημαντικότερο ρόλο και μεταξύ άλλων και ελέγχου, νομικού ελέγχου και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα ενισχυθεί αναλόγως. Η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων έγινε πια δεσμευτική, παραδείγματο χάρη. Υπάρχει λοιπόν τώρα πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη ισορροπία, εξισορρόπηση μεταξύ σεβασμού δικαιωμάτων και αποτελεσματικότητας. Όταν προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε και να συνδυάσουμε την πολιτική δίωξη του εγκλήματος, βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά στον ακαδημαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα αυτά που βλέπετε εδώ, το Corpus Juris του 97 και τον οικονομικό νόμο της Ένωσης, του οποίου, τον οποίο επιμελήθηκε ο καθηγητής Τίμερμαν. Τέλος, το μανιφέστο για την Ευρωπαϊκή Ποινική Πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι, για να το πω έτσι, έχουμε μια καλή βάση πια για να συζητήσουμε την εγκληματολογική ή ποινική πολιτική της Ευρώπης γιατί έχουμε αυτή τη συνθήκη πως τη λένε της Λεσαβόνας και η τελευταία σχετική δήλωση της Κομισιόν είναι αυτή που θα σχολιάσω γιατί ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ακριβώς να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Uh, Σε αυτή την ανακοίνωση της Κομισιόν δίνεται μια βάση για μια πιο συνεπή ποινική πολιτική της Ένωσης και η δυνατότητα οι βασικές αυτές αρχές να καθοδηγούν το σύνολο της ποινικής νομοθεσίας της Ένωσης. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, λέγω. Οι βασικές αρχές που βλέπετε εδώ δικαίως αναφέρονται από την ανακοίνωση της Κομισιόν, δηλαδή η αρχή της επικουρικότητας, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αναγκαιότητα αναλογικότητας και τέλος η ultima ratio. Και στην εφαρμογή των διώξεων και στον καθορισμό των κυρώσεων είναι σημαντικά αυτά τα κριτήρια. Ε, και βέβαια η αρχή της νομιμότητος είναι σημαντική. Πολύ βασική, Όταν συγκρίνουμε την ανακοίνωση αυτή της Κομισιόν με το μανιφέστο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Δίωξη του Εγκλήματος, που κατήρτισαν ακαδημαϊκοί βλέπουμε ότι βλέπουμε σε ποιο σημείο η απέτηση να υπάρχει θεμητός και νόμιμος στόχος ως τμήμα της Ultima Ratio είναι πολύ σημαντική. Στο μανιφέστο αυτό λοιπόν τονίζεται ιδιαίτερα αυτή η αρχή Και στα δύο έγγραφα όμως, οι αρχές, ultima ratio, αναλογικότητα, επικουρικότητα κλπ. δεν περιγράφονται σε μεγάλη λεπτομέρεια και ένα από τα κυριότερα καθήκοντά μας για το μέλλον θα ήταν ακριβώς να δούμε με πιο συνοπτικό, πιο πλήρη τρόπο τι σημαίνουν οι αρχές αυτές και ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος τους. Συζητιέται πολύ στους ακαδημαϊκούς κύκλους η Ultima Ratio. Αλλά το περιεχόμενο της είναι ακόμη ασαφές. Σας είπα τι λέει ο βόρειος συνάδελφός μου που βλέπετε εδώ για τη χρήση του ποινικού δικαίου κ. Άλμποργ είναι μία αρχή που καλύπτει θα έλεγα όλες τις υπόλοιπες και δεν πρέπει να την ξεχνάμε όταν συζητάμε το μέλλον του ποινικού δικαίου στην Ένωση. Το θέμα της ποινική αξίας σχετίζεται προφανώς για παράδειγμα με το θέμα αυτό του θεμητού ή νόμιμου στόχου η αρχή της χρησιμότητος ή η σύγκριση του ωφέλους επίσης σχετίζεται και η αρχή της ανθρωπιάς καθώς και η αρχή της φρόνησης, δηλαδή της χρησιμοποίησης όσο το δυνατόν λιγότερων νομικών ποινικών μέσων. Σε ενωσιακό επίπεδο, η αρχή της Ultima Ratio σχετίζεται άμεσα με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βασίζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στα δύο αυτά έγγραφα την ανακοίνωση της Επιτροπής και το Μανιφέστο γίνεται παραπομπή σε αυτή την αρχή γιατί και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ζητάει τον περιορισμό της χρήσης ποινικών διώξεων στο ελάχιστο δυνατόν, στο απαραίτητο. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία ιδιαιτερότητα του ποινικού δικαίου είναι ότι οι διώξεις δημιουργούν και κοινωνικό στιγματισμό και ηθική ταπείνωση. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα του ποινικού δικαίου σε σύγκριση με άλλα δίκαια. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον καθορισμό των βασικών αρχών που πρέπει να το διέπουν, διότι το δικαστικό ποινικό σύστημα πρέπει να εμπνευστεί από αυτές τις αρχές. Το πρόβλημα της δημοκρατικής νομιμότητας και της εμπιστοσύνης προς το σύστημα είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί. Και πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα και εμπιστοσύνη. Επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που είπαμε στην αρχή. Οι αρχές της ultima ratio, επικορικότητα και αναλογικότητα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Συμφωνώ με αυτά που λέει το μανιφέστο ότι τα επιχειρήματα περί νομιμότητος πρέπει να συνοδεύουν τη συνέπεια του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και άρα τίθεται το ερώτημα τι θα ήταν αυτή η συνέπεια. Αυτό συζητήθηκε και στο προηγούμενο γύρο βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει να καταφέρουμε να πετύχουμε τη συνέπεια του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου αλλά ταυτόχρονα ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια εναρμόνιση του, των εθνικών ποινικών δικαίων γιατί και αυτό θα ήταν μεγαλύτερη συνέπεια. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος υπερβολικής διαφοροποίησης, δηλαδή να δημιουργηθούν δύο είδη συνέπειας ευρωπαϊκού επίπεδου στο οικονομικό επίπεδο και μετά στο ποινικό. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα για την εφαρμογή της αρχής της Ultima Ratio. Το λέει και το μανιφέστο. Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο επιχειρημάτων που προκύπτουν από το προγενές δικαίω της Ένωσης, τα συντάγματα των χωρών μελών και της χάρτας των θεμελιωδών. ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία ενωσιακού επίπεδου διώξεων σε ποινικό επίπεδο. Τα είπε και ο καθηγητής Κλιπ. Αλλά μπορεί τα κριτήρια που αναφέρονται εδώ και που προκύπτουν από το πρωτογενές δίκαιο να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν ιδιαίτερα για τον οικονομικό ποινικό δίκαιο. Ορισμένοι λένε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν ρήτρε σε επενωσιακό επίπεδο και άλλοι όχι. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα της νέας ρήτρα στο άρθρο 83.2 που μας δίνει τεράστιες δυνατότητες συζήτησης του κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιείται το ποινικό δίκαιο ως μέσον. Αλλά είναι και αυτό μια βάση, μια βάση για να ζητήσουμε να απαιτήσουμε την εφαρμογή του κριτηρίου του θεμελιώδους συμφέροντος. Αυτό δεν αρκεί βέβαια. Αρκεί. Πρέπει να γίνουν και περισσότερες, πιο λεπτομερείς διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή των κριτηρίων αναλογικότητας, επικουρικότητας. και υπάρχει και αυτή η δοκιμή που βλέπετε εδώ αναγκαιότητο ή μη της εφαρμογής ενωσιακού ποινικού δικαίου το βλέπετε εδώ ανάποδα για μας η αρχή της αναλογικότητας και επικουρικότητας συνδέονται βέβαια συνδέονται. εδώ σας λέω ποιες είναι οι βασικές συνταγματικές ή νομικές ρήτρες στη συνθήκη της Ένωσης και στο πρωτόκολλο εφαρμογής των. Και υπάρχει και αυτό το σημαντικό άρθρο στο 83.3 Emergency Break. Οι αρχές αυτές πρέπει να είναι βέβαια νομικά δεσμευτικές και τα κριτήρια για την αξιολόγηση και χρήση τους και εφαρμογή τους δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Κάποτε πρέπει να γίνει και αυτή η επεξεργασία γιατί γιατί δεν υπάρχει νομολογία για τη χρήση αυτού του, στις της αρχής της επικουρικότητας, ενώ υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και μπορεί να σας αναφέρω μετά και μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν δύο-τρεις αποφάσεις που έχουν μεγάλη σημασία. Συνήθως γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας από τη μία και των πραγματικών νομικών επιπτώσεων από την άλλη. Η επικουρικότητα θα πει αν η Ένωση πρέπει να παρέμβει και η αναλογικότητα πώς να παρέμβει. Αλλά συνδέονται φυσικά. Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται κυρίως για την επίλυση διαφορών μεταξύ ατόμων ή μεταξύ πολιτών και δημοσίου και υποδιαιρείται σε τρεις υποκατηγορίες κατά πόσον είναι κατάλληλη η αρχή αυτή, κατά πόσον είναι απαραίτητη και κατά πόσον είναι αναλογική στρίκτο σένσου. Αυτέ Αυτές είναι οι βασικές απλώς κατανομές και διαχωρισμοί και χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για να αναπτυχθεί η εφαρμογή των αρχών αυτών στο μέλλον της ποινικής πολιτικής της Ένωσης. Ε, λοιπόν, για να σεβαστώ και το χρόνο μου θα φτάσω στα συμπεράσματα. Τα έχετε ξανακούσει αυτά που λέει εδώ, ανάποδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο μέλλον στο μέλλον. Τέτοιου είδους αναλύσεις θα χρειάζονται όλο και περισσότερο αξιολογήσεις, προτάσεις, συγκρίσεις εφαρμογών συγκεκριμένων περιπτώσεων στα ποινικά δίκαια και επίσης πολύ περισσότερη έρευνα με βάση συγκεκριμένες περιπτώσεις ως βάση που να αποτελέσουν τη βάση μιας πιο εξορθολογισμένης Δίωξη του εγκλήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα προκλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της, όπου δεν υπάρχει και τόσο συνομολογία. Και ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι αξιολογήσεις, ανεξάρτητες μάλιστα. Όπως είπατε και στο προηγούμενο γύρο σας, κατευχαριστώ. Εμείς σας κατευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας γιατί δεν έχουμε επαρκή. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο κύριος ε, <clears throat> Ζάτσκερ, ε, καθηγητής ε, ποινικού δικαίου, οικονομικού ποινικού δικαίου και ποινικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και τον παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεγιόγκ ε, και την ε, πρόεδρο που οργάνωσε αυτή τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως είπατε <clears throat> είναι πολύ κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλη εξουσία για την κατεύθυνση της πορείας της αντιμετωπίσεως του ποινικού δικαίου στο μέλλον. Ε, θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο μου θέμα για να μην επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη λεχθεί στο θέμα της νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ιδίως κατά την μεταφορά <coughs> της νομοθεσίας στον εθνικό τομέα. Ε, θα, από την αρχή θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι θα αναφερθώ στον γερμανικό ποινικό κώδικα που ανέρχεται στο 1935 την εποχή των Ναζί και έλεγε ότι ε, όποια πράξη θεωρείται αξιόπινη από την νομοθεσία ή ε, αντιτίθεται στο ε, ο <clears throat> λαϊκό αίσθημα θα τιμωρείται διότι για μένα η αρχή αυτή είναι πολύ καλή εισαγωγή διότι μας δίδει μία εγγύηση δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά μας αποδεικνύει και την πρακτική σημασία. Θα χωρίσω την ομιλία μου σε τέσσερα θέματα. Καταρχήν την νομοθεσία αυτή καθεαυτή. Ε, δεύτερο, τη σημασία της ε, νομικής ε, συμμαχίας και την εφαρμογή της και γιατί οι νομοθέτες πρέπει να αναφερθούν, να αναφέρονται ή στην νομική νομοθεσία και τι προτείνω για να υπάρξει βελτίωση η αρχή της νομιμότητας σήμερα δεν είναι μόνο θέμα δικαίου το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη αλλά ένα διεθνώς αναγνωρισμένο διεθνές δίκαιο και τα περισσότερα συντάγματα αναφέρονται στο θέμα αυτό όπως άλλωστε και ο νέος χάρτης που αναφέρεται στην αρχή της νομιμότητας την οποία μπορούμε να καθορίσουμε σαν νούλουμ κρίμεν νούλαμ πένα. Εάν δεν υπάρχει έγκλημα δεν υπάρχει και κύρωση δηλαδή. Και βλέπουμε ότι όλες αυτές οι αρχές είχαν καταστρατηγηθεί από την πρώην ναζιστική ρύθμιση και ε, βλέπουμε ότι η εφαρμογή αυτή είναι εις βάρος του δράστη και δεν εξασφαλίζει νομική βεβαιότητα, λέξ σέρτα. Ε, και ε, θεωρούμε ότι αυτά τα σημεία είναι στο επίκεντρο του θέματος που θα αναπτύξω σήμερα διότι το άτομο πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει ε, τι πράξεις ή τι ελλείψεις τον οδήγησαν εις το να διώκεται. Η αρχή της νομιμότητας λοιπόν πρέπει να είναι αμοιβαία όταν εφαρμόζεται ο ποινικό κώδικας αλλά εάν αντιλαμβανόμαστε την ποινική νομοθεσία σαν τη γερμανική υπάρχει μία ερμηνεία και ε, σημαίνει ότι ε, δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά ποινικά δικήματα ούτε ο ευρωπαϊκό ποινικό δικαστήριο. Και μόνο εάν υπάρχει αρμοδιότης ε, να ε, υπερκεραστεί ε, η εθνική νομοθεσία μπορεί να επιτρέψει εφαρμογή ευρωπαϊκών διατάξεων που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση δεν είναι πολύ σαφής όταν μιλάμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου ελέγχθησαν, ε, όπως ελέγχθη ε, ήδη ε, στο άρθρο 335 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον στη θεωρία θα μπορούσε να νομοθετήσει για την πάταξη των ποινικών οικονομικών εγκλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει τον όρο της European Fraud αλλά αυτό είναι κάτι που παραμένει για το μέλλον και άρα ο νομοθέτης προς το παρόν δεσμεύεται πλήρως από την νομιμότητα. Όλοι πρέπει να μπορούν να προβλέψουν ε, γιατί θα ευθύνονται και να υπάρχουν και αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια ε, και ένα ε, προβλέψιμο σύστημα κυρώσεων και ένα γνωστό σύστημα ερμηνείας των αδικημάτων. Οπότε ε, δεν ε, μπορεί να υπάρξει μία απόφαση στο τέλος, αλλά θα πρέπει για όλα τα αδικήματα τα οποία αποτελούν ευρωπαϊκά αδικήματα να υπάρξει κάποια υποδομή και ε, ένα νομικό πλαίσιο των Ευρωπαίων νόμων νομοθετών που θα έχουν καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό ποινικό ε, δίκαιο. Ε, λόγω του ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ποινικών ε, δικαίων σε εθνικό επίπεδο θα υπάρξουν και μεγάλες αντιδράσεις σε ένα τέτοιο εγχείρημα και τώρα θα επανέλθω στα ουσιαστικά μας προβλήματα δηλαδή πώς μπορούμε να καταρτήσουμε ζητήσουμε μέτρα που θα εναρμονίζουν την νομοθεσία των κρατών μελών όπου η νομιμότητα αμφισβητείται. Άρα πρέπει να αναλύσουμε ε, πολύ προσεκτικά τις δυνατότητες. Ποια είναι η, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Καταρχήν αναφέρομαι εις την συνθήκη σύμφωνα με την οποία μπορεί ο νομοθέτης να καταρτήσει ένα πλαίσιο ο, ελαχίστων κυρώσεων. Επειδή μιλάμε για εναρμόνιση και για καθοδήγηση των εθνικών νομοθετών. Δεν ξέρω αν αυτό συμβιβάζεται με ευρωπαϊκή νομική βεβαιότητα. Και σύμφωνα με τον ορισμό στις συνθήκες ε, θα ε, δεσμεύουν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις στα κράτη-μέλη αλλά ε, δεν θα τις δεσμεύουν δεσμεύουν πέραν του να νομοθετήσουν σε εθνικό επίπεδο επί των θεμάτων αυτών. Γιατί λοιπόν θα συμμορφωθούν οι εθνικοί νομοθέτες εάν ε, μπορούν να προβλέψουν ένα σύστημα το οποίο θα προκαθορίζει τις ευθύνες και τις ποινές τότε που είναι το πρόβλημα. Ε, φέτος, ε, έχει δημοσιευθεί στις αρχές του χρόνου ένα σχετικό έγγραφο όπου προβλέπεται ότι η εθνική και υπερεθνική νομοθεσία δεν επηρεάζεται πάντοτε στο ίδιο επίπεδο αλλά είναι ε, κάπως ε, πολύ ανυπεύθυνο να θεωρήσουμε ότι οι εθνικοί νομοθέτες πάντοτε πρέπει να διορθώνουν το θέμα της ε, των ευρωπαϊκών αποφάσεων σχετικά με την ε, ε, νομική ασφάλεια διότι εδώ υπάρχουν δύο αρχές το δικαίω, το, υποχρέωση νομιμότητος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών και το, την υποχρέωση να υπάρχει νομική βεβαιότητα στο άρθρο 4 της οδηγίας προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να υπάρξουν τουλάχιστον κυρώσεις 10 ετών φυλάκισης για άτομα που διακινούν άλλους ανθρώπους και ο εθνικός όμως τις μπορεί να πει ε, εάν μιλάμε για φυσιολογικές ή σοβαρές αξιόπινες πράξεις πώς θα τις διαχωρίσουμε και μεταξύ τους και ε, από τις πολύ σοβαρές αξιόπινες πράξεις. Οπότε ε, μπορεί να γίνει μία, ε, μία διατύπωση η οποία θα είναι απλώς πιο σαφής από αυτήν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και για τις για ε, ε, τη, ρύθμιση αυτή θα μπορούσε στη Γερμανία ε, το σοβαρό αδίκημα, ποινικό αδίκημα να προσωμιαστεί με αυτό το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 26 του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα. Για να υπάρχει όμως προβλεψιμότητα στο εθνικό ποινικό σύστημα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση ο εθνικός νομοθέτης και υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές οι οποίες ε, αν ερμηνευθούν ευρέως μπορεί να θεωρηθούν σαν υποχρεώνοντας να εφαρμόσει κανείς μία οδηγία υπό προϋποθέσεις που δεν καλύπτονται από την εθνική νομοθεσία. Δηλαδή μία μείωση της ακοής κατά 50% μπορεί να θεωρηθεί ως όχι αρκετά σοβαρή βλαβή σε εθνικό επίπεδο ενώ εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίσει ότι αυτή η βλάβη είναι πολύ σοβαρή θα καταδικάσει το κράτος ε, για μη πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Άρα αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη στο θέμα της ε, βεβαιότητος της νομιμότητος και ε, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η νομική βεβαιότης. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη κατά κάποιον τρόπο να εξασφαλίσουν συμπληρωματική βεβαιότητα και αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής. Όσο λιγότερο είναι το λάθος στην εφαρμογή, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει εξασφαλίσει την αρχή της λέξης σέρτα και αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στο ποινικό δίκαιο. Με το ίδιο παράδειγμα, αν το κράτος δεν μπορεί να ε, εφαρμόσει και να ερμηνεύσει την σοβαρή βλάβη τότε θα πρέπει να υπάρξει μία ελάχιστη διατύπωση η οποία να καθοδηγεί τους εθνικούς νομοθέτες. Ε, όταν λοιπόν ε, να αρμονίζουμε την νομοθεσία ε, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτά τα θέματα αλλά μπορούμε να παραπέμψουμε και σε άλλες ε, νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παραδείγματος χάρη για την προστασία του περιβάλλοντος και την κάλυψη της προστασίας αυτής από, τη, από το ποινικό δίκαιο όπου ο εθνικός νομοθέτης θα πρέπει να νομοθετήσει χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εθνική νομοθεσία και αυτό είναι εις βάρος της νομικής βεβαιότητας της πράξεως και πρέπει να διευκρινίζουμε και να διαχωρίζουμε την νόμιμη από την παράνομη πράξη και αυτό δεν είναι δυνατόν υπό αυτές τις συνθήκες και τα εθνικά ποινικά δικαστήρια πρέπει να εφαρμόζουν αυτή την νομοθεσία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να υπάρξει ένας περιορισμός σε αυτή την τεχνική, δηλαδή ο νομοθέτης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ε, ε, νομική βεβαιότητα σε όλο το εύρος ε, του εγχειρήματο διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο απέδειξε ο κύριος Κλίνκ ότι δηλαδή θα είναι αδύνατο να υπάρξει μία καταδίκη. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ε, λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα και τέλος μπορούμε να δημιουργήσουμε ποινικό δίκαιο υψηλού επίπεδου και κατόπιν της συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κατάλληλο σημείο για να αναλυφθεί αυτή η ευθύνη για την εξέλιξη του ποινικού δικαίου διαφορετικά όλα τα συστήματα απλώς θα καλύπτουν την προληπτική λειτουργία τους. Εάν είμαστε συνεκτικοί μεταξύ ε, ευρωπαϊκού και νομικού και εθνικού ποινικού δικαίου θα μπορέσουμε πολύ καλύτερα να σεβαστούμε την νομιμότητα θα υπάρξουν διατάξεις οι οποίες θα προβλέπονται εις οδηγίες και στη συνέχεια και σε κανονισμούς και θα μπορέσει σε κάποιο σημείο να υπάρξει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ε, ποινικό δίκαιο. Χρειάζεται λοιπόν η συνεκτικότητα, η συνοχή ε, και όλες οι αρχές θα πρέπει να διατηρούνται ε, και να υπάρχει μία υποχρεωτική ε, διαβούλευση όταν ε, χειριζόμαστε θέματα ποινικού δικαίου και αυτό πρέπει να συζητηθεί μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον κάποια στιγμή ε, να υπάρξουν ορισμένες εμπειρίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστεί ε, ένα απόθεμα εμπειρίας με το οποίο θα συνεργάζονται και διεθνείς ομάδες ε, παραδείγματος χάρη η ε, πρωτοβουλία η ομάδα που ε, έκανε τη διακήρυξη μπορεί να αξιολογήσει τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο μανιφέστο και θα αποτελεί μια καλή βάση συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζον Σπέσερ που είναι καθηγητής νομικής στο Πανεπιστημίο του Κέμπριτζ ε, και κατόπιν θα έχουμε μια πάρα πολύ σύντομη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Ντε ε, που μας κάλεσε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Είναι τιμή μου που με προσκαλέσατε σε θέματα ποινικού δικαίου και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου είμαι ρασιτέχνης. Εγώ είμαι καθηγητής ε, στο αγγλικό ποινικό δικαίο και στην ε, αγγλική δικονομία και να σας πω ως ιστορικό ότι ουσιαστικά στα μάτια πολλών συμπατριωτών μου είμαι κάτι σαν ερεκτικός, γιατί ήμουν τμήμα της ομάδας ε, που συνέταξε το Project Corpus Euros και ουσιαστικά κυκλοφόρησε την ιδέα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Και αυτή ε, η ιδέα ουσιαστικά ερμηνεύτηκε ως ε, συνωμοσία των Βρυξελών για να αντικατασταθεί το common με το Ναπολεονικό σύστημα και όπως ε, ορισμένοι μπορεί να γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο ε, στη χώρα μου πέρασε μια νομοθεσία για να καταστήσει πιο δύσκολο για το Ηνωμένο Βασίλειο να ακυρώνει αλλαγές στη συνθήκη απαιτώντα δημοψήφισμα πριν να μπορέσουμε να ακυρώσουμε διάφορα μέτρα που αφορούν και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Και νομίζω ότι μεταξύ των ακαδημαϊκών νομικών αυτό μου δίνει μία μοναδική διάκριση. Πολλοί ακαδημαϊκοί είχαν ιδέες που απορρίφθηκαν Νομίζω ότι πρέπει να είμαι ο μόνος ε, που συνέβαλε στο να ε, κυκλοφορήσει μια ιδέα που θεωρήθηκε ότι ήταν τόσο τρομερή που τροποποιήθηκε το σύνταγμα της χώρας έτσι ώστε να γίνει σίγουρο ότι ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτή στο μέλλον. Μια πιο ήπια εκδοχή της ε, αντίστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο είναι η έννοια ότι το σύστημα common law κατά κάποιο τρόπο δεν είναι συμβατό με το ποινικό δίκαιο ε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου και ότι επομένως εφόσον είναι ασύμβατο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο ενέο σύστημα που θα ταιριάζει και στους δύο. Αυτή φυσικά δεν είναι η δική μου οπτική. Εγώ δεν πιστεύω ούτε καν ότι αληθεύει κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά τις ποινικές διαδικασίες και σίγουρα δεν ισχύει σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο που είναι το αντικείμενο της ακρόασης αυτής. Και στους νομικούς ε, της Ευρώπης έλεγαν, ε, ποτέ, έλεγαν συχνά ε, οι νομικοί του Common Law ότι το Common Law δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί και βασίζεται σε προηγούμενο. Και φυσικά αυτό διαφέρει κάπως από το σύνορο στην υπηρετική Ευρώπη που έχετε κώδικες. Αν αυτό ίσχυε κάποτε, δεν ισχύει σήμερα, δεν αληθεύει σήμερα. Σήμερα τα περισσότερα ποινικά δικήματα στην Αγγλία και στην Ουαλία βασίζονται και προσδιορίζονται από το νόμο, από το statute και είναι αλήθεια ότι εξακολουθούμε να έχουμε αντικείμενα common law, δηλαδή που δεν βασίζονται σε νομική βάση και εξαρτώνται αποκλειστικά σε ε, δικαστικό προηγούμενο, κάτι που εφευρέθηκε από τους δικαστές πριν χρόνια λέγοντας «Α, αυτό είναι κακό, είναι είναι έγκλημα» βάσει του άρθρου 2 του Γερμανική Νομοθεσίας του 1935, στο οποίο αναφέρθηκε πριν λίγο ο κύριο ε, Ζάτσκερ, ο καθηγητή Ζάτσκερ, αλλά οι δικαστέ μα πλέον ε, δεν ισχυρίζονται ότι έχουν την αρμοδιότητα να αναπτύξουν ε, το ποινικό δικαίωμα δηλώνοντα νέα αδικήματα. Έχουν τελειώσει αυτέ οι μέρε, έχουν τελειώσει αυτέ οι εποχέ των δικαιωμάτων common law και σιγά σιγά αντικαθιστώνται αυτά τα δικήματα από δικήματα που βασίζονται στο νόμο, στο τέτοιο το Και ε, σχεδόν όλος ο ε, κόσμος του common law βασίζεται τώρα σε ποινικού κώδικες, σε πλήρες ποινικού κώδικες. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο συνέταξε κώδικες ποινικού και στην εποχή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και στα περισσότερα μέρη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας είχαν ε, ουσιαστικά νομοθεσία που κωδικοποιήθηκε. Και τελικά κάναμε εξαγωγές, αλλά ποτέ δεν ε, καταναλώθηκαν ε, στο ίδιο το εσωτερικό. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι κατορθώνουμε να επιβιώσουμε κάποια δυσκολία χωρίς να έχουμε τέτοιες κώδικες, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι κάπως πολύπλοκο. Η απουσία ποινικού κώδικα σημαίνει ότι υπάρχει διαφορά μορφής μεταξύ του ποινικού δικαίου στι δικές ε, νήσους ε, και στις χώρε τη υπηρετική Ευρώπη. αλλά σε ό,τι αφορά στην ουσία νομίζω ότι υπάρχει πολύ μικρή πραγματική διαφορά σε ό,τι αφορά το γενικό τμήμα του ποινικού δικαίου, οι κανόνες που σχετίζονται με το στοιχείο της ενοχής, με τα ποινικά δικαιώματα, οι κανόνες που σχετίζονται με την ενοχή, με την α, παρότρινση, τη συνωμοσία και την απόπειρα και με ε, τη γενική περάσπιση. Σε όλους αυτούς τους κανόνες δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ε, επί των αρχών που να διαχωρίζουν το common law με τον κόσμο της υπηρετικής Ευρώπης και τέτοιες διαφορές, ε, αν υπάρχουν, νομίζω ότι δεν είναι μεγαλύτερες από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορών νομικών συστημάτων στο εσωτερικό ε, της Υπηρετική Ευρώπης. Και το ίδιο νομίζω ισχύει ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή ε, των αδικημάτων μιλώντα Εβραίου, οι ίδιοι κακοί άνθρωποι, δηλαδή, μπορεί να τιμωρηθούν για τι ίδιε κακέ πράξει, ανεξάρτητα με το αν ε, έχουν ε, διαπράξει το αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Υπηρετική Ευρώπη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει γέννη διαφορά μεταξύ του κόσμου, του common law και τη Υπηρετική Ευρώπη ε, σε ό,τι αφορά αυτό που αποκαλούν οι Γάλλοι η ποινική πολιτική, la politique penale, δηλαδή τις αρχές βάσει τις οποίες ε, οι νομοθετές αποφασίζουν ποια συμπεριφορά θα ποινικοποιείται στο μέλλον. Και στον κόσμο του common law, όπως και αλλού, οι θεωρητικοί φαίνεται να επιχειρηματολογούν ε, ότι η ποινική νομοθεσία πρέπει να είναι ultima ratio, το έσκατο μέσο, αλλά οι κυβερνήσεις και μάλιστα πρόσφατα έχουν τίνει έχουν την τάση να δημιουργούν νέα αδικήματα και χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο προτεραιοτήτων. Τα πρώτα δεκαέτη της εξουσία των εργατικών που εκλέχθηκαν το 1997 λέγεται ότι περίπου 3.000 νέα αδικήματα δημιουργήθηκαν. Και κάποιοι κοινικοί λένε, στην, την διαφράση όπως είπε και ο Κορνίλης Δεγιόγκ, ότι οι πολιτικοί τείνουν να δημιουργούν νέα ποινικά δικήματα ως ένα φτηνό και εύκολο τρόπο να φαίνεται να κάνουν κάτι για ένα πρόβλημα ε, και δίνουν μια απάντηση την οποία κανείς δεν καταλαβαίνει. Αν ρωτήσετε μένα και αν μου πείτε να ονομάσω, να κατονομήσω τις ε, προφανείς διαφορές μεταξύ του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στην Αγγλία και στην Ουαλία, το τμήμα δηλαδή του κοικομολόγου που ξέρω καλύτερα και του ουσιαστικού ποινικού δικαίου ε, στα κράτη της Υπηρετικής Ευρώπης που γνωρίζω, θα έλεγα ότι γενικά οι κύριες διαφορές είναι ότι ο δικό μας ε, νόμος τίνει να είναι πιο αυστηρός. Τα μεμονωμένα δικήματα τείνουν να, να καθορίζονται ευρύτερα, δηλαδή ε, παραδείγματο χάρη αν έχουμε ε, κάποια ε, επίθεση και δολοφονία. Είναι πολύ πιο ευρία η έννοια αυτή από όσο γνωρίζω. Επίσης, είμαστε πολύ πιο ικανοποιημένοι να δημιουργούμε κάποια δικήματα που αφορούν την αμέλεια ε, και την ευθύνη από τις άλλες χώρες ε, και την, υπάρχει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογή ε, για την υπεράσπιση και οι μέγιστες ποινές φαίνεται να είναι υψηλότερες. Περνούν χάρη 7 χρόνια για την απλή κλοπή. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό. Κάποιος ε, μου έθεσε αυτήν την ερώτηση κάποτε και είπα ότι πιθανότατα γιατί οι κανόνες μας, ε, οι δικονομικοί κανόνες που έχουμε, καθιστούν τόσο δύσκολο να συλλάβουμε κάποιον, έτσι λοιπόν όταν το συλλαμβάνουμε τον χτυπάμε πολύ σκληρά. Και έτσι λοιπόν το σύστημά μας είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και βαρύ και ε, υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στοιχεία διακριτικέ ευχέρειας. το χάρη ο εισαγγελέα δρά ε, στα πλαίσια τη ευκαιρία του να ασκήσει δίωξη, σε αντίθεση με άλλε χώρε, Ιταλία, Γερμανία, όπου υπερισχύει αρχή τη νομιμότητα. Δεύτερον, έχουμε ε, την ε, ε, jury equity, δηλαδή ε, η ισότητα των ενόρκων, παραδείγματο χάρη όταν έχουμε κακουργήματα, ε, συμμετέχουν και οι ένορκοι ως δικαστές και μπορούν να αθώσουν και ουσιαστικά αυτό λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα κατά της ε, πολύ αυστηρής νομοθεσίας και επίση τα δικαστήριά μας έχουν πολύ μεγάλη ευχαίρεια ως προς την επιβολή ποινών. Έτσι λοιπόν ε, η άποψη ότι το ουσιαστικό δίκαιο στις χώρες του Common Law ε, διαφέρει τόσο πολύ από το ουσιαστικό δίκαιο στις ε, χώρες της υπηρετικής Ευρώπης ε, είναι τόσο μεγάλη που σήμαινε ότι οι Βρυξέλλες δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ποινικό δίκαιο, δεν ισχύει. Αν οι Βρυξέλλες προσπαθούσαν του χάρη να μειώσουν τις μέγιστες ποινές, κάτι τέτοιο θα έρχονταν σε αντίθεση με τα κυρία χαρακτηριστικά του ποινικού δικαίου σε όλα τα σήμερα, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή είναι μια εξέλιξη, πιθανή εξέλιξη στην Ευρώπη. Ακούγοντας ε, τους υπόλοιπους ομιλητές σήμερα το πρωί, αναρωτήθηκα Υπάρχει κάποιο γενικό μάθημα που μπορεί να σας δώσει το Ηνωμένο Βασίλειο όταν ε, ζητούμε το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι ίσως ε, υπάρχει. Στο Ενωμένο Βασίλειο Έχουμε τρία διαφορετικά νομικά συστήματα, Αγγλία και Ουαλία, Σκοτία, Βόρεια Ιρλανδία και στο επίπεδο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου έχουμε κάποιες ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών. Παραδείγματος χάρη η έκτορση είναι σχεδόν ε, παράνομη στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ είναι διαδέσιμη κατόπιν αιτήματος ε, δυνάμει της νομοθεσίας Αγγλίας και Σκοτίας. Επίσης, η ηλικία σεξουαλικής συνένεσης είναι στα 17 στη Βορεια Ιρλανδία, ενώ είναι 16 σε άλλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και όταν υλοποίησαμε το καθήκον μας να εφαρμόσουμε την πρώτη οδηγία για την εμπορία ανθρώπων, στο... Ε, υπήρχαν διαφορές ε, στο δίκαιο της Αγγλίας από το δίκαιο της Σκοτίας, ε, αλλά παρόλα αυτά μπορέσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς μεγάλες διαφορές και αν αυτό μπορεί να γίνει στο εσωτερικό μιας χώρας, από ό,τι φαίνεται, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ φυσικά συμφωνώ ε, με τον συνάδελφο Αντρικλίπ για την αναγκαιότητα του να έχουμε υπερβολικά εναρμονισμένο, υπερβολικά πολύ εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή ουσιαστικά ε, αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματο σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την αμοιβή αναγνώριση. Εμεί λειτουργούμε τρία συστήματα με κάποιε διαφορέ ουσιαστικού ποινικού δικαίου βάσει τη αμοιβή αναγνώριση των αποφάσεων του δικαστηρίου και νομίζω ότι αυτό ήταν το μάθημα που έδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν δική μα ιδέα που υιοθετήθηκε για να περάσουμε στην αμοιβή αναγνώριση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει, επομένω θα κάνουμε μια πολύ σύντομη συζήτηση. Βλέπω ότι ο Σάρμπερ θέλει να θέσει κάποιε ερωτήσει. Σα παρακαλώ σε ένα λεπτό, αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει έχω. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Η πρώτη είναι σχετικά με την αρμοδιότητα εναρμόνισης του ποινικού δικαίου αυτή τη στιγμή. Εργαζόμαστε τώρα επί διατάξεων για την ε, καταπολέμηση του κλίματος στον κυβερνοχώρο, εργαζόμαστε για την εναρμόνιση των ε, διατάξεων του ποινικού δικαίου. Και μερικές φορές δεν είναι σαφές που υπάρχει σύνδεση με τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων. Και φαίνεται να υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το πώς θα προσδιορίσουμε αυτές τις διατάξεις ποινικού δικαίου. Και ακούσαμε κάτι από τον κύριο Ζάτσκερ ότι πρέπει να είμαστε ακριβείς όταν ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά α, βάσει της δικής μου εμπειρία δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα μέχρι τώρα. Και δεύτερη ερώτηση. Αν ε, εναρμονίζουμε το ποινικό δίκαιο, φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένε προκλήσεις. Και αναρωτιέμαι, αν θα συμφωνούσατε ότι σε ορισμένου τομεί ε, περισσότερο έχουμε να κάνουμε με πρόληψη παρά με εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που θέλω να θέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία λόπε και μετά θα απαντήσουν οι πανελιστές. Μάλιστα, όπως είπε Κάλμπρεχ, στη δική μας ε, περίπτωση πολλές φορές ε, εκπονούμε νομοθεσία για την πρόληψη και εδώ έχουμε δυσκολία. Παραδείγματο χαρή, ε, εισηγήτρια για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία για να προστατεύσουμε τις γυναίκες ε, που είναι αντικείμενο κρατικών μεταχείρισης. Και τα προβλήματα που βλέπουμε είναι ότι ο ορισμός ε, του αδικήματος άσκησης βίας κατά των γυναικών δεν είναι ίδιος ε, στα κράτη-μέλη. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα δεν ορίζεται αυτό το δίκημα. Και καθώς εδώ έγινε αναφορά στο ότι πρέπει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια ε, Το τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για βία καθώς ε, προφέρουμε στην εκπόνηση προληπτικής νομοθεσίας, βρισκόμαστε σε, μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί όταν ένας δικαστής ε, ή μια διοικητική αρχή εκτιμούν ότι πρέπει να εκδώσουν εντολή προστασίας επειδή υπάρχει αυτή η απειλή και μέχρι ποιο βαθμό θεωρείται απειλή που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών. Αυτή ήταν μια συζήτηση που αφορούσε και τις διάφορες ε, νομικές παραδόσεις των χωρών, γιατί σε κάποιες χώρες την εντολή αυτή την εκδίδουν αστυνομικές αρχές, ε, σε άλλες χώρες διοικητικές αρχές και σε άλλες δικαστές. Έτσι λοιπόν εγώ θέλω να ρωτήσω. Εμείς πιστεύουμε εδώ ότι είναι λογικό να πάμε μέχρι και έναν ορισμό του αδικήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν ορίζεται το αδίκημα και το Συμβούλιο της Ευρώπης ήδη έχει συνάψει μια σύμβαση ορίζοντας το αδίκημα και διευκρινίζοντας σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών. Γιατί βρισκόμαστε στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων. Και στο παρελθόν δεν έχουμε συναντήσει αυτή τη δυσκολία. Ήθελα λοιπόν να μου πούν οι ακαδημαϊκοί την άποψή τους για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Κάρμεν. Έχουμε και τον εκπρόσωπο της ε, Low Society, της ε, Ένωσης ε, Νομικής. Προερχόμαι από την... Ναι, είμαι από την νομική εταιρεία Αγγλίας-Ουαλίας. Η ερώτησή μου αφορά και τον προηγούμενο γύρο και αυτόν. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στο μέλλον στο εξής. Αν αυτές οι σημαντικότατες αποφάσεις ληφθούν στο ενωσιακό επίπεδο, δηλαδή κατά πόσον επιβάλλεται η δημιουργία ενός ενωσιακού ποινικού δικαίου ή κατά πόσον πρέπει να εναρμονιστούν τα ποινικά δίκαια των χωρών μελών, τότε τι ρόλο βλέπουν οι ομιλητές για τους νομομαθείς, για τους επαγγελματίες σε αυτή τη φάση αν θέλουμε να καθορίσουμε τι πολιτική θα οδηγήσει τις αποφάσεις αυτές, ποιος είναι ο ρόλος των νομικών σε αυτή την πρώιμη φάση για τα πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απαντήσουν οι ομιλητές. Ορίστε, αρχίστε εσείς. Καλά, ας αρχίσω εγώ αφού δεν θέλουν οι άλλοι. Λοιπόν, θα απαντήσω με τη σειρά των ερωτήσεων. Κύριε το θέμα ήταν νομίζω διπλό. Ποιε ακριβώ είναι οι δικαιοδοσίε και δεύτερον ποιε είναι οι νομικέ πράξεις. Οι δικαιοδοσίες βασίζονται στις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι συνθήκες. Με... Στη Γερμανία γνωρίζουμε ότι το συνταγματικό δικαστήριο είναι πάντοτε πολύ ακριβές και Δεν νομίζω ότι θα ήταν παράλογο να πούμε ότι βασιζόμαστε στις συνθήκες και πρέπει να οδηγούμαστε από τις συνθήκες. Εκεί θα δούμε αν η συνθήκη μας δίνει καμία δικαιοδοσία οποιοδήποτε είδους. Να ερμηνεύσουμε λοιπόν τις συνθήκες για να δούμε αν οι προτάσεις που γίνονται μπορεί να θεωρηθεί ότι βασίζονται σε αυτές. Επίσης, μιλήσατε για την αναγκαιότητα ή μη αντιμετώπισης των εγκλημάτων με ενωσιακό τρόπο. Πρέπει και εδώ να υπάρξει λεπτομερέστερος ορισμός στις οδηγίες. Γιατί εδώ θα αρχίσει να εφαρμόζεται η αρχή της νομιμότητας και η πιθανή εναρμόνιση της νομοθεσίας. Είπατε κάτι σημαντικό, ότι η πρόληψη είναι σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη από ότι η κύρωση, η τιμωρία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να συμπεριλαμβάνεται σε οποιαδήποτε αξιολόγηση πρώτα να δούμε αν η πρόληψη είναι δυνατή και με τι εργαλεία και μόνο αν αυτό δεν λειτουργήσει να προχωρήσουμε στις κυρώσεις. Αυτή είναι η βασική ιδέα του Ultima Ratio. κυρία Ρομέρο Λόπες, μιλήσατε για την κακομεταχείριση των γυναικών. αν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κάποιο είδους συμπεριφορές πρέπει ακόμα μια φορά να έχουμε πρώτα καλύτερους ορισμούς για να γνωρίζουμε ποιες ακριβώς διοκτικές αρχές εφαρμόζονται στην κάθε περίπτωση. Τέλος, δεν θυμάμαι το όνομα της κυρίας στο τέλος, από την νομική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πολύ χρήσιμο χρήσιμη η εμπειρία των νομικών και νομομαθών για να μας πούν και εκείνοι είναι αποτελεσματική η τιμωρία των αδικούντων. Όχι μόνο οι ακαδημαϊκοί και οι καθηγητές που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και οι νομικοί γενικά πρέπει να μας δώσουν τη συμβουλή τους. όλοι οι ασχολούμενοι με τον νόμο να γνωμοδοτήσουν για το κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ενωσιακό ποινικό δίκαιο. Σας κατευχαριστούμε κύριος Λάχτη τώρα. Απλώς θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι ε, υπέρ του να ε, χρησιμοποιήσει κανείς την εμπειρία των σκανδιναβικών χωρών που έχουν ε, ένα μεγάλο απόθεμα και εξετάζουν σφαιρικά το θέμα της πολιτικής, της ποινικής πολιτικής <clears throat> αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής ποινική πολιτικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, ε, ποινικής οικονομίας. Όσον αφορά το άρθρο 83.1, νομίζω ότι η αρχή της επικουρικότητας, παραδείγματος χάρη, πρέπει να ε, λαμβάνεται υπόψη και όταν έχουμε ασαφείς ε, ορισμούς θα πρέπει να τους κοιτάξουμε πάρα πολύ λεπτομερώς διότι οι αρχές αυτές είναι ε, πάρα πολύ ευρείες και θα πρέπει να υπάρξουν επιπρόσθετα επιχειρήματα σχετικά με το ultima ratio. Οπότε ε, βάσει του άρθρου 83 αυτές είναι οι σκέψεις που μπορούμε να αναπτύξουμε ε, σχετικά με το άρθρο 85 ε, και όταν μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις Πρέπει ε, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε διότι προς το παρόν είναι πολύ ασαφής η αντιμετώπιση. Δεν έχω να σας προσθέσω κάτι συγκεκριμένο σχετικά με την πρώτη ερώτηση αλλά όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα με εντυπωσίασε ότι η βία ε, κατά των γυναικών ε, είναι νόμιμη σε ορισμένα κράτη-μέλη και αντιλαμβάνουμε ότι ένα τέτοιο ο κράτος ε, ε, θα ε, καταδικαστεί είτε από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη είτε γενικότερα όσον αφορά την συμμετοχή των πρακτικών στο θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και την ώρα που μιλούσε η ερωτούσα να ποιος είναι ο μηχανισμός που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και μπορεί να βελτιωθεί διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σε οργανισμός που ονομάζεται Φόρουμ Δικαιοσύνης και μπορεί εκεί να συζητήσει ε, κανείς διάφορες ιδέες διότι υπάρχουν νομικοί οποίοι εξασκούν το ε, τομέα, το επάγγελμα ε, και Διεπίστωσα ότι κατόπιν πρωτοβουλίας του κυρίου Ντιάντζελης που ήταν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου επειδή εγώ ήμουν ομόλογος του για το ε, ε, Ηνωμένο Βασίλειο και είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος περιλαμβάνει επαγγελματίες από διάφορους τομείς προσπαθούσαμε να απαντήσουμε σε ερωτηματολόγια και να προωθήσουμε ορισμένες συζητήσεις και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πολλές φορές αναλαμβάνει έρευνες και ε, εξετάζει διάφορα θέματα ε, ερωτώντας τους επαγγελματίες και εγώ έχω υπάρξει εισηγητής για τέτοια θέματα ρωτάει αν ο μηχανισμός αυτός αρκεί και ε, αν όντως μπορεί να προχωρήσει. ότι ε, θα πρέπει ε, να ε, εξετάσει κανείς τα άτομα που εξασκούν το επάγγελμα τι χρήζει βελτιώσεως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια αυτά και τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε και να καλέσω το, την τρίτη στρογγυλή τράπεζα ευχαριστώντας προηγουμένως τους συνομιλητές μου σε αυτό το χώρο Ε, thank you very much. I would like... Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω τα μέλη του πάνελ και θα ήθελα να περιοριστείτε στα 10 λεπτά αν είναι δυνατόν προκειμένου να έχουμε και λίγο χρόνο στο τέλος ε, για να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Λοιπόν, ε, πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Λότε Κνούτσεν, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο και να μας συνοψίσετε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Λυπή και τον κύριο Τεγιόγκ για την ευκαιρία να μιλήσουμε σε αυτή την ακρόση για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για το ποινικό δίκαιο. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και νομίζω ότι αυτό μας δείχνει ε, πόσο επίκαιρο είναι το ζήτημα σήμερα που βρισκόμαστε σχεδόν δύο έτη μετά τη θέση ισχύ της Λισαβόνας και αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τη συνθήκη και να βιώνουμε μια νέα περίοδο για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Θέλω να καλύψω δύο θέματα. Καταρχήν την ανακοίνωση μου, την ανακοίνωση μας, με συγχωρείτε, του Σεπτεμβρίου σε σχέση με την ε, ε, πολιτική ποινικού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών τη Ένωση μέσα στο ποινικό δικαίου και πώ θα έχουμε συνοχή στην χάραξη τη ποινική νομοθεσία. Με την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, η Κομισιόν ε, για πρώτη φορά ανέφερε την άποψή τη σε σχέση με ένα σύνολο αρχών που διέπουν ε, την νομοθεσία στο ποινικό τομέα από το νέο νομικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι οι νέε ευκαιρίε ε, που προσφέρονται από τη Λισαβόνα αποτελούν ευκαιρία να ξεπεράσουμε μια σειρά ελλείψεων και κατακαιρματισμών τη νομοθεσία που ξέραμε από τον τρίτο πυλώνα και να εισαγάγουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Η καταπολέμηση του εγκλήματο είναι ένα από του τομεί ε, όπου νομίζω αναμένεται πράγματι μεγαλύτερη δράση. Είναι ένα από τα θέματα που τονίστηκαν ε, και στην έκθεση Αλφάνο. Αλλά επίση γνωρίζουμε ότι το common ε, law ε, είναι ε, ουσιαστικά ένα πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα με ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην προσέγγιση μας γιατί το ποινικό δίκαιο είναι ένας τομέας ε, όπου η ποικιλομορφία στην Ευρώπη μεταξύ των κρατών μελών είναι μεγάλη και δεν νομίζω ότι σε κανέναν άλλο τομέα του δικαίου αντικατοπτρίζονται εκεί πολύ περισσότερο τα ήθη και τα έθιμα των κοινωνιών και παραδόσεις και η συνθήκη της Λισαβόνας δέχεται και προστατεύει αυτή την ποικιλομορφία των νομικών συστημάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 62. Και για το λόγο αυτό Χρειαζόμαστε σαφείς και διαφανείς κανόνες για το πότε χρησιμοποιούμε το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Το νομικό μας ε, πλαίσιο έχει αλλάξει σημαντικά από τη Συνδίκη της Λισαβόνας. Αναφερθήκατε ήδη στη μετάβαση στην απόφαση. Ε, κυρίως έχουμε το νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ισότιμος παίκτη στην νομοθετική διαδικασία και φυσικά έχουμε και το δικαστικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά ακόμη και με αυτές τις αλλαγές συνθήκη η βάση παραμένει ίδια Μιλάμε για το σεβασμό του εισαρχή τη επικουρικότητα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπω αναφέρονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες ε, που να μπορούν να οδηγήσουν στη ελευθερία και γι' αυτό η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει τα όρια για τη δράση μας ε, η χάρτα είναι υπό την ευθύνη της Αντιπρόεδρου Ρέντινγκ που είναι αρμόδια και για δικαιοσύνη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι υπάρχει μια ισχυρή λογική στο να συνδυάσουμε στον ίδιο φάκελο αυτές τις δύο συνιστώσεις ε, γιατί η χάρτα φαίνεται ε, να παρουσιάσει το σπιξίδα για τις πολιτικές μας ε, και μας παρέχει τον πυρήνα των κανόνων για την προστασία των πολιτών και φυσικά πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη για το ποινικό δίκαιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ ε, επικεντρώνεται η ανακοίνωση στο άρθρο 83.2 που πρώτη φορά αποτελεί μία ε, βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης ε, και φυσικά οι αρχές διέπουν το ευρύτερο πλαίσιο του ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ήδη είχαμε ένα προηγούμενο πριν τη Λισαβόνα με δύο οδηγίες για περιβαλλοντικό δίκαιο και την ρήπαση της θάλασσας 2008-2009. Αυτά ήταν τα πρώτα νομοθετήματα που εφετήθηκαν ε, στο ποινικό δίκαιο με διαδικασία συναπόφασης και βασίστηκαν σε πολύ καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο τότε. Και αυτές οι δύο οδηγίες μέχρι τώρα θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν μελετά την μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο από τα κράτη-μέλη για να δει αν υπάρχει αναγκαιότητα follow-up. Στην ανακοίνωσή μας εμείς προτείναμε μία προσέγγιση σε δύο στάδια και όπως είπε κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές, ίσως να μην είναι τόσο λεπτομερής, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια. Πρώτη φορά εμείς, οποιοδήποτε άλλο όργανο, ε, νομίζω ότι συγκέντρωσαν όλα αυτά σε ένα και μόνο έγγραφο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η αρχή και η διτή προσέγγιση μας ε, παρέχει μια βασική μεθοδολογία πώς θα καθορίσουμε τα κατόφλια που πρέπει να ισχύουν ε, για την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι κατευθυντήριες αρχές είναι η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα και η επικουρικότητα και κυρώσει του ποινικού δικαίου φυσικά επιβάλλονται για τα πολύ σοβαρά δικήματα ε, και φυσικά πάντοτε μιλάμε για σκατομέσο όταν χρησιμοποιούμε το ποινικό δίκαιο. Η συνθήκη ε, έχει το δικό της τεστ και της δοκιμή ρωτώντα αν είναι ουσιαστικά τα μέτρα ποινικού δικαίου για να πετύχουμε αποτελεσματική εφαρμογή τη πολιτική. Και αυτή είναι ουσιαστικά η ουσία και αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτη θα πρέπει να αναλύσει αν υπάρχουν άλλα είδη κυρώσεων διοικητικών λόγου χάρη που μπορεί να μας ικανοποιήσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια της επιβολής. Και αν ε, τελικά υπάρχει ανάγκη ποινικού δικαίου, υπάρχει δεύτερο βήμα που πρέπει να εξετάσουμε τι είδου μέτρα ποινικού δικαίου πρέπει να φοιτήσουμε και εδώ συνθήκη θέτει τα δικά τη όρια, γιατί περιορίζει τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ελάχιστου κανόνε για τον ορισμό των αδικημάτων και των κυρώσεων που φυσικά καλύπτουν την αρχή της νομιμότητας, ε, όπως ε, ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Και πάλι, οι αρχές της αναλογικότητας ε, και της αναγκαιότητας θέτουν επίσης όρια σε σχέση με το είδος των ποινικών κυρώσεων και το επίπεδό τους. Και τέλος, ε, χρειαζόμαστε κάποια στατιστικά στοιχεία για να θεσπίσουμε τους κανόνες ε, και πληροφορίες για τις ε, αποκλήσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, τον αντίκτυπο στις κυρώσεις και το πιθανό έλλειμμα στην επιβολή. Το θέμα του ελλείμματος επιβολής είναι πολύ σημαντικό καθώς οι ποινικέ κυρώσει μπορούν να αποτελούν ένα στοιχείο ενδυνάμισης ε, της πολιτικής επιβολής νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν ε, την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποφασίζουν από μόνα τους συνήθως πώς θα το πράξουν αυτό. Ω προ την επιβολή, αλλά το ποινικό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να προβλέψει, να παρέχει ένα πρόσθετο εργαλείο για την εφαρμογή των πολιτικών τη Ένωση και ε, ε, ε, ποιες άλλες πολιτικές, σε ποιε άλλε πολιτικέ μπορούμε να έχουμε ποινικά μέτρα, μέτρα ποινικού δικαίου. το ορισμένε εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε ότι η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να ενδυναμώσει τι πολιτικέ σε ε, επιλεγμένες συναρμονισμένου ε, επιλεγμένους συναρμονισμένους τομείς και αυτό θα γίνεται με αξιολόγηση αναπερίπτωση των ε, διάφορων κενών στην εφαρμογή. Θέλω να αναφέρω όμως τρία παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων που νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα σχετικά στη σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο, οικονομικό πλαίσιο, προστασία του χρηματοοικονομικού τομέα καταρχήν και όπως αναφέρθηκε η Κομισιόν τον Οκτώβριο εκπώνησε μια πρόταση οδηγία για ποινικέ κυρώσει για το insider dealing και για την χειραγώγηση τη αγορά που αποτελούν τμήμα ενό ευρύτερου πακέτου για να αντιμετωπίσουμε τι ελλείψει στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεύτερον, έχουμε το θέμα τη απάτη, όπω αναφέρθηκε από πολλού ομιλητέ η απάτη συγκεκριμένα που θίγει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί επικεντρωνόμαστε και σχεδιάζουμε την υποβολή μια πρόταση το 2012 για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που θα καλύπτουν τα κενά που έχουμε από τη Σύμβεση του 1995 για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τρίτον, να αναφέρω την προστασία του ευρώ κατά της παραχάραξης και κυβδηλίας. Αυτός είναι ένας τομέας επίσης στον οποίο θα παρουσιάσουμε νομοθεσία του χρόνου προκειμένου να ενδυναμώσουμε τη συνολική εμπιστοσύνη στα μέσα πληρωμών. Υπάρχουν καλοί εναρμονισμένοι τομεί πολιτική, όπου το ποινικό δίκαιο εν θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για την επιβολή όμως όλα αυτά τα μέτρα θα πετούσαν ε, πολύ περαιτέρω ενέλυση και εξέταση πριν ε, να πάμε παραπέρα. Υπάρχουν κάποια παράδειγμα που αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας βέβαια. Και να πω και δύο λόγια για κάποιες ε, θεσμικές πτυχές ή κάποιες μεθόδους εργασίας που αναφέρθηκαν εδώ μεγαλύτερη σαφήνεια και συνεκτικότητα είναι ένας από τους κύριους στόχους μας και νομίζω ότι το ε, η ίδια η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ δικαιοσύνη διευκόλυνε αυτή η διαδικασία σε επίπεδο κομισιών, γιατί κατά πολλού τρόπου εμεί παρέχουμε μία πύλη, αν θέλετε, με δεξοδό για άλλε τομεικέ υπηρεσίε ε, που θα ήθελαν ε, να εξετάσουν τη λήψη μέτρων ποινικού δικαίου δυνάμει του 83.2. Μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπαθίες μας, να παρέχουμε συμβουλές και διδάγματα. Έτσι λοιπόν, εσωτερικά εμείς ως Κομισιόν προσπαθούμε να διασφαλίσουμε συνοχή και συνεκτικότητα σε ε, ε, επίπεδο υπηρεσιών και η ΓΑΜΑ Δικαιοσύνη ε, διασφαλίζει ότι υπάρχουν διάφορες εξελίξεις στον τομέα του ποινικού δικαίου για τη λήψη νέων μέτρων και προβαίνουν σε έγκαιρη περιοδοποίηση για οποιαδήποτε σχέδια για μέτρα ποινικού δικαίου σε άλλους τομείς και επίσης εμείς προσφέρουμε υποστήριξη και αρρωγή αν σκοπεύουν να κάνουν περαιτέρω εξέταση του ποινικού δικαίου και αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι είναι συνεκτική όλη η διαδικασία ακόμη και πριν την ε, σχεδιασμένη αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το φόρουμ για τον εσωτερικό συντονισμό. Επίσης, ε, πέρα από τις προτάσεις μας, προετοιμάσαμε, προετοιμάζουμε, με συγχωρείτε, και μελέτες αντικτύπου, δηλαδή αιτιολογού, εξετάζουμε αν αιτιολογείται ε, η πρόταση και τις διάφορες επιλογές πολιτικής, όπως και την επιλογή που έχουμε κάνει. Και αυτές οι μελέτες αντικτύπου θα αντιμετωπίσουν πολλές από τις ερωτήσεις ε, και τα θέματα που τέθηκαν και έχουν να κάνουν με την επικορικότητα, την αλογικότητα και άλλες βασικές αρχές. Και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση στο μέλλον ε, θα αφήσει κάποιο ανεξίδηλο σημάδι στις ε, προτάσεις μας ε, για το ποινικό δίκαιο. Και είπαμε και στην ανακοίνωσή μας και το επαναλάβαμε πολλάκις ότι είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε πραγματικά αποδεκτικά στοιχεία. Για κάθε μία από τις προτάσεις μας πρέπει να τονίζουμε ποια είναι η λογική και ποιο είναι το αποτέλεσμα και πρέπει αυτό να το υποστηρίζουμε με πραγματικά γεγονότα, με στατικά στοιχεία, ε, των νομικών συστημάτων των κρατών μελών σε συγκριτική βάση. Πρέπει να αναλύουμε ε, τον αντίκτυπο στην νομοθεσία, την υφισταμένη κατάσταση στα κράτη-μέλη, ποιες είναι πώς οι διαφορές στα διάφορα καθεστώτα επιβολής κυρώσεων μπορεί να έχουν ε, ε, τον τάδι αντίκτυπο τελικά. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλές εξελίξεις, ε, προσπαθούμε ουσιαστικά να έχουμε μια πρόταση η οποία βασίζεται σε αποδείξεις και ταυτόχρονα η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, δικαιοσύνης ε, εξετάζει και τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά καταρτίζουμε ένα ε, είδος καταλόγου, checklist, κάνουμε έναν έλεγχο ποιότητας και παρακολουθούμε και τη μεταφορά της νομοθεσίας στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών. Αυτό είναι ουσιαστικό καθήκον. Και ήδη να οργανώνουμε εργαστήρια για να το κάνουμε αυτό ή κάποια προγράμματα. Έχουμε το Γιουλίτα, παραδείγματο χάρη, ε, όπου ε, το, ε, ασχολούμαστε με τις προσπάθειες της μεταφοράς και της εφαρμογής της ροποθεσίας για την παροχή διερμηνίας και μετάφρασης. και Έχουμε και μια διαδικασία τριών σταδίων, όπου έχουμε συστήματα με συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και εργαστήρια. Έχουμε ένα σταδίο παρακολούθησης, ε, reporting, υποβολή εκθέσεων. Και έχουμε και ένα στάδιο επιβολής. Ε, αναφέρω τις οδηγίες ε, για την ρήπαση στη θάλασσα πριν το σχάρι, γιατί εκεί πρώτη φορά παρακολουθούμε την εφαρμογή με τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία κατά παράβαση. Και επίση ε, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να απτύξουμε περαιτέρω τον προβληματισμό του ποινικού δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το ανακοινώσαμε στην ανακοίνωσή μα και ελπίζουμε ότι αυτή η ομάδα θα αρχίσει να λειτουργεί το 2012 και θα μα βοηθήσει να διερευνήσουμε νομικά ζητήματα. Υπάρχει μια σειρά νομικών ζητημάτων που πρέπει να διερευνηθούν και να εξεταστούν όπως ε, και θέματα όπως ε, ο σύνδεσμος μεταξύ διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ίσως και να ερμηνεύσουμε νομικές έννοιες όπως παραδείγματος χάρη παραόντρηση, υποβοήθηση. Το ή σημαίνουν οι αποτελεσματικέ, αναλογικέ και αποτρεπτικέ κυρώσει. Έχουμε μία σειρά πραγμάτων εδώ που μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και πρέπει να διερευνήσουμε λεπτομερώς. Και ένα από τα άλλα θέματα αυτές της ακρόασης ήταν η ποιότητα της νομοθεσίας. Νομίζω είναι ένας τρόπος να πούμε ποιότητα της δικαιοσύνη. γιατί όπως τονίστηκε, ε, οι δικαστές χρειάζονται ε, ακρίβεια και ασφάλεια δικαίου στους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν με ένα σωστό και ομοιόμορφο τρόπο. Έχουμε υπερβολική ευελιξία στην ερμηνεία και νομίζω ότι αυτό μας ε, καθοδηγεί και στην νομοθετική διαδικασία και είναι επίσης σημαντικό για τα κράτη-μέλη που πρέπει να μεταφέρουν στο δίκαιό τους μια οδηγία και χρειάζονται να γνωρίζουν καλύτερα ποιο είναι ο στόχος και ποια είναι η πρόθεση μιας συγκεκριμένης διάταξης. Να αναφέρω και κάτι ακόμα σε ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν σχεδιάζουμε διάφορες μελέτες, δύο μελέτες για το περιβαλλοντικό δικαίο και για τη ρήπα στη θάλασσα. Γιατί αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε εδώ, για να εξετάσουμε το σύστημα των κυριώσεων στα κράτη-μέλη και να συγκρίνουμε την κατάσταση και να απαντήσουμε σε κάποιες ανησυχίες που ακούστηκαν. Έτσι λοιπόν πολλά περισσότερα θα κάνουμε ως ε, προς ε, την ε, διοργάνωση μελετών και συντονισμού προσπαθειών. Θέλω λοιπόν συμπεριέτω να πω ότι όλα αυτά μας έδειξαν πώς η Κομισιόν μπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ε, ποινικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι μια συνεκτική τέτοια πολιτική μπορεί να φέρει προσθεμένη αξία για την καταπολέμηση του βίου εγκλήματος και να απαντήσουμε σε ανησυχίες των πολιτών και στην αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. Το ποινικό δίκαιο αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερη έννοιας του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνη, που αφορά και την αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ δικαστικών αρχών στις διάφορες χώρες, καθώς και τους ελέγξητους κανόνες ε, για τα δικονομικά δικαιώματα, στις ποινικές διαδικασίες, καθώς και για τα θύματα. Και, για να τελειώσω, Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αναπτύξουμε μια κοινή κατανόηση πολλών ε, των καθηγητηρίων αρχών που διαπούν το ποινικό δίκαιο και γι' αυτό καλωσορίζουμε τις προσπάθειες του κ. Ντεγιόγκ και τη επιτροπή ΛΥΜΠΕ να διερευνήσει τις έννοιες αυτές. Ε, πραγματικά ευπρόσδεκτη η συνεισφορά σας και φυσικά αυτά θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα, σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριος ε, Τόμας Οστροπόλσκι. Έχετε το λόγο. Thank you very much, and good morning everyone, and thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα τον κύριο Ντεγιόγκ για την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε να μιλήσουμε εξ ονόματος της Πολωνικής Προεδρίας και μάλιστα του Συμβουλίου. Διότι πράγματι μια συνεπής προσέγγιση στο ποινικό δίκαιο πάντοτε θεωρούνταν σημαντική από το Συμβούλιο. Μου ζήτησαν εδώ να μιλήσω για τις ρήτρες που προβλέπονται για, στο εξή για το ποινικό δίκαιο, αλλά πριν το κάνω αυτό θα ήθελα σύντομα να περιγράψω με το ιστορικό από το 2 και μετά. Μόλις τέθηκε ενισχύ δηλαδή η συνθήκη της Λισαβόνας για να δούμε τουλάχιστον λίγο πώς προσπάθησε το Συμβούλιο να προσεγγίσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Ήταν πολλά και είχαν πολλές διαστάσεις. ιδιοκτικές διαδικασίες, οι αλλά και άλλα θέματα και άλλα που θα τα αναφέρω στα απλά μου, στις απλές μου διαφάνειες. Λοιπόν, το δύο, το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του, σε συμπεράσματα του, πράγμα που δεν ήταν τυχαίο γιατί ήταν μόλις αμέσως η ενισχύει της συνθήκης, ανέφερε ορισμένες καινοτομίες, ε, καινοτομίες στον τομέα του ποινικού δικαίου στην Ένωση. Ίσως να γνωρίζετε ότι η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου ήταν πολύ περιορισμένη μόνο σε ορισμούς εγκλημάτων. Ακόμη και τώρα οι συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ποινικό δίκαιο δεν υπησέρχονται στο θέμα των κυρώσεων. Ακόμα και συμβάσεις για τη δουλεμπορία δεν, ακόμη και του 11, δεν θέτουν το θέμα των κυρώσεων. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ήταν το πρώτο βήμα τότε το 2. Μόλις άρχισε να ισχύει δηλαδή η συνθήκη της Λισαβόνας γιατί τότε κατάλαβαν τα κράτη-μέλη συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν νέα προβλήματα και νέα πρόκληση προς αντιμετώπιση. Ενώ ταυτόχρονα ήθελαν να διατηρήσουν την ελαστικότητα και το περιθώριο ελιγμών των. Χρειάστηκε βέβαια κάποια συνέπεια, αυτό είχε αναγνωριστεί και τα δύο κύρια στοιχεία της προσέγγισης του Συμβουλίου ήταν να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της μελλοντικής νομοθεσίας για το ποινικό δίκαιο για να δούμε αν η εφαρμογή αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων θα ήταν αποτελεσματική ή όχι ή μήπως δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί να εφαρμοστούν συγκεκριμένες και αυστηρές κυρώσεις αναλογικά βέβαια. Στα συμπεράσματα εκείνα του 2 που αποτελούν τη βάση των μελλοντικών αναλύσεων, που αποτέλεσαν τη βάση των μελλοντικών αναλύσεων, προστέθηκε μία σημαντική παρατήρηση, δηλαδή ότι ένα σημαντικός όρος ότι δεν πρέπει τίποτα να εμποδίσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν κατώτατα όρια κυρώσεων όπως εκείνα θεωρούσαν ότι έπρεπε να επιβληθούν. Αυτή ήταν η αρχή λοιπόν. Αυτή ήταν η αρχή και το επόμενο βήμα έγινε το 6 μετά από τις αξιοσημείωτες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την μόλυνση όπου το δικαστήριο ακύρωσε ορισμένες εθνικές αποφάσεις λέγοντας ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις και πέρα από τον τρίτο πυλώνα. και ότι μπορούν οι ποινικές, ρήτρε να αποτελέσουν πλέον τμήμα ενωσιακών νομοθετικών εργαλείων. Αυτό βέβαια δημιουργούσε τον κίνδυνο κάποιας ασάφειας γιατί, ή ασυνέπειας γιατί αν στην περίπτωση που τέτοιου είδους ποινικέ ρήτρες είχαν αναπτυχθεί εκτός της γνωμοδοσίας των ειδικών, τότε, τότε λέγω δημιουργούνταν μια φοβερή ασάφεια. Γι' αυτό προβλέφθηκε όλες οι αποφάσεις με, οι νομοθεσίες με ποινικέ ρήτρες να υποβάλλονται στην ομάδα εργασίας για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο που γνωμοδότησε για τέτοιες ρήτρες από πολύ νωρίς για να υπάρχει να διασφαλίζεται κάποια συνέπεια, νομική συνέπεια. Αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέρθηκε το Συμβούλιο για το θέμα. Τέλος, τέλος. Μου ζητήθηκε να περιγράψω ένα άλλο εγγραφό. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ποινικό δίκαιο του 5. Ο τίτλος τους λέει κατευθυντήριες γραμμές για, το ποινικό δί... για την προσέγγιση του Συμβουλίου προς το ποινικό δίκαιο. Ήδη από τη συνθήκη της Λισαβόνας είχε αποσαφινιστεί ότι θα έχει νέο ρόλο το ποινικό δίκαιο ακόμη και στα πλαίσια της ενωσιακής πολιτικής της κατάρτισης των ενωσιακών προγραμμάτων. Για το Συμβούλιο λοιπόν θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό να αποφανθεί για τις κατευθύνσεις τις οποίες έπρεπε να κινηθεί και να αναπτυχθεί το ποινικό δίκαιο. και τονίστηκαν τρία ωφέλη που θα είχε αυτό. Να γίνουν διαπραγματεύσεις ως προς την ουσία των ποινικών ρητρών, διευκόλυνση της μεταφοράς του στο εθνικό δίκαιο, ερμηνεία τους εθνικά αν προηγουμένως είχαν βασιστεί, αν είχαν βασιστεί σε προηγούμενα νομικά στοιχεία και κατευθυντήριες γραμμές. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εκείνα έχουν δύο τμήματα, το δεξί και το αριστερό. Το πρώτο αφορά γενικές αρχές της εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Το έχουν πει και άλλοι προηγουμένως και Κατά το Συμβούλιο το ποινικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται μόνον, μόνον σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για ultima ratio. Φυσικά με αναλογικότητα και επικουρικότητα δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ αυτά. Τέλος, τονίστηκε ότι η προστιθέμενη αξία των ποινικών ρητρών πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί πριν αποφασιστεί να εφαρμόζεται συστηματικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο λόγω της μεταβλητής γεωμετρίας που ισχύει πια στο Συμβούλιο. Γιατί μόνο 24 κράτη αντί 27 συμμετέχουν στην ε, δημιουργία αυτών των ε, εργαλείων ποινικού δικαίου. Αντίθετα από το 6 όπου είχε ζητηθεί να συμμετάσχουν όλα τα κράτη. Ορισμένα σημαντικά στοιχεία που αναφέρουν αυτά τα συμπεράσματα δείχνουν πώς ακριβώς το Συμβούλιο βλέπει τις ποινικέ ρήτρε που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Αυτά που γράφω εδώ. Για τις κυρώσεις υπόθηκε ότι έπρεπε να συμφωνούν με τα συμπεράσματα του 2002. ή τουλάχιστον να μην αντιφάσκουν αν και μπορούσαν να τα ξεπεράσουν. Θυμηθείτε και τι είπε προηγουμένως η κυρία Λούτιφορντ. Ε, αυτές οι δηλώσεις ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν ε, <coughs> για να ε, προωθήσουν και να βοηθήσουν στις συζητήσεις στο Συμβούλιο και θα αποτελέσουν μόνο ένα σημείο ενάρξεως για να μπορέσουν να βελτιωθούν και οι περαιτέρω εξελίξεις οι οποίες έτσι θα είναι πιο συγκεκριμένες. Και τέλος χρειάζεται μία εποπτεία αυτών των διατάξεων αλλά το Συμβούλιο στην αρχή ήταν μάλλον επιφυλακτικό διότι θεώρησε ότι αυτή η λύση θα ήταν ε, γραφειοκρατική για να δημιουργηθεί μία επιπλέον τεχνολογία. Εξού και ε, στη συνέχεια και το Συμβούλιο, οι γραμματείες ε, και οι υπηρεσίες θα λάβουν υπόψη αυτές τις διατάξεις. Μέχρι στιγμής όμως τα προβλήματα αυτά δεν έχουν προκύψει στην πρακτική ε, παρόλο που είπα ότι υπάρχουν και άλλα θέματα και ε, όλα αυτά δεν είναι στο επίπεδο των συγχρόνων διατάξεων τις οποίες θα ελπίζαμε αλλά ε, νομίζω ότι σε ορισμένα από αυτά τα θέματα ιδίως σε ένα υπάρχει μία μονάδα η οποία παρακολουθεί την νομοθετική ακρίβεια των διαφόρων κειμένων τα οποία προβλέπονται κατά τρόπον ώστε κάθε Υπουργείο να μπορέσει να παρουσιάσει το θέμα. Θα σταματήσω λοιπόν τώρα, με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η διερμηνία πρέπει να απελευθερωθεί. Υπάρχει ακόμη ένας ομιλητής, οπότε ε, ο κύριος Αντώνιο Κραγιόλα, ο οποίος ήταν, ε, είναι ο επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. Κύριε ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να παρουσιάσω ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορεί δηλαδή η νομική υπηρεσία να βοηθήσει ε, καλύτερα την Επιτροπή Ελευθεριών σε θέματα νομικής και ποινική διαδικασίας διότι υπάρχει μία παράδοση ότι πολλές αρχές πολλές φορές ε, αλλάζουν από γλώσσα σε γλώσσα και ερμηνεύονται διαφορετικά και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη παρόλο που συνήθως όπως ξέρετε ε, κινούμαστε ε, στα γαλλικά και αγγλικά σαν σαν γλώσσες εργασίας. Υπάρχουν όμως ορισμένες διαδικασίες ε, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη και θα ήθελα να αναφερθώ εις ε, τα πρώτα ε, βήματα το δικαίωμα να υπάρχει διερμηνία στις, στις ποινικέ διαδικασίες και το θέμα του ε, ουσιαστικού δικαίου σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να ακολουθηθεί μία διαδικασία όπου θα υπάρχει διαβούλευση ε, με την νομική υπηρεσία και αυτό έχει ε, αποφασιστεί από το Προεδρείο το Ιανουάριο του 2004 και μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να υπογράψουν και να υποβάλουν ένα γραπτό το ερώτημα για νομική γνωμοδότηση και εγώ μπορώ εδώ ε, να βασιστώ στην εμπειρία μου εις ε, την σύνδρομη σε διάφορες ε, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των οποίων θα μπορούσα να αναφέρω την Επιτροπή Ελευθεριών, την Επιτροπή Αραφορών κτλ. Εδώ ασχολούμεθα με πάρα πολλά θέματα μεγάλη σημασίας και όπου έχουμε ε, ασχοληθεί ε, τις ε, προηγούμενες χρονιές και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε το φόρτο εργασίας του Κοινοβουλίου και έχουμε προσπαθήσει να έχουμε γραπτές νομικές γνωμοδοτήσεις ε, κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να συνδράμουμε ιδίω στην Επιτροπή Ελευθεριών και βλέπουμε ότι πολλές φορές στήθενται ενδιαφέροντα καινοτόμα ερωτήματα στην ε, νομική υπηρεσία χωρίς να υπάρχει επαρκής χρόνος να τα εμβαθύνουμε για προφανείς λόγους γιατί τίποτα δεν είναι προφανές όταν πρόκειται για καινοτόμα θέματα ή ευαίσθητα θέματα όπως είναι θέματα του Σέγγεν ή θέματα της ε, διαμόρφωσης μιας ποινική πολιτικής. Επίσης ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν απαντούμε μόνο σε γραπτά ερωτήματα αλλά και σε προφορικά ερωτήματα επιτόπου, πράγμα το οποίο είναι μεγάλη πρόκληση για το προσωπικό της υπηρεσίας μας, κατά τρόπον ώστε να είμαστε επικοδομητικοί και πρέπει να σας πω ότι η μονάδα μας που ασχολείται και με ποινικά θέματα παρακολουθεί όλες τις ε, διαδικασίες για να έχει ε, πέντε σημειώματα για κάθε διαδικασία σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή όπου γίνεται μία νομική ανάλυση ε, βάσει της ε, ε, προτάσεως που έχει υποβληθεί σχετικά με την διαδικασία την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε και ουσιαστικές αρχές όπως είναι η επικουρικότητα, τα θαμελιώδη δικαιώματα και ε, τον ε, υποκείμενο ποινικό, το υποκείμενο ποινικό δίκαιο. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν συμμετοχή στις συνεδριάσεις που οργανώνονται από τον εισηγητή και στους τριμερείς διαλόγους μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Είναι λοιπόν μία ουσιαστική νομική βοήθεια και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι η νομική υπηρεσία είναι εξοπλισμένη κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, υπάρξει σεβασμός του ποινικού δικαίου αλλά οι υπηρεσίες μας πολλές φορές δεν έχουν επαρκές δυναμικό κατά τρόπον ώστε να μπορούν να παρακολουθούν εφόλης τη θέματα και ε, πρέπει να ασχοληθούν και με άλλα θέματα δικαστική συνεργασία, άσυλο, Σένιεν και τα θέματα εκεί είναι πολύ διαφορετικά από τα θέματα που τίθενται στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να κάνουμε μία, έναν διαχωρισμό μεταξύ της ε, ποινική δικονομίας και των άλλων θεμάτων. Χρειάζεται εξειδίκευση και χρειάζεται να έχει κανείς κατάλληλα άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί συγκεκριμένα και έχουμε ήδη αυτό το προσωπικό πράγμα το οποίο επιτρέπει ίσους δικηγόρους και νομικούς μας να εμβαθύνουν διάφορα διάφορα θέματα, ιδίω όταν είναι πολύ εξειδικευμένα, όπως παραδείγματο χάρη τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να υπάρχει μία μόνιμη επαφή με τους συναδέλφους της ε, γραμματείας ΛΥΜΠΕ κατά τρόπον ώστε να μπορεί ε, προχωρήσει πιο αποτελεσματικά. Θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει και μία ε, παρακολούθηση της βοηθείας στις επιτροπές και να υπάρχει μία μόνιμη επαφή με τους συναδέλφους οι οποίοι ε, εξετάζουν την ε, ε, ποινική δικαιοσύνη και την ποινική δικαιονομία, πράγμα το οποίο απαιτεί εξαιρετική γνώση των ποινικών δικαίων των 27 χωρών και μία ενημέρωση συνεχή και παρακολούθηση του ισχύοντος συστήματος ποινικού δικαίου διότι διαφορετικά τα έγγραφα που παρουσιάζουμε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι ε, ε, νομικές γνωμοδοτήσεις σύμφωνα με το πνεύμα του κανονισμού 1049 στην περίπτωση Τούρκο παραδείγματος χάρη. Οπότε παρόλα αυτά ε, είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για να συνδράμουμε ιδίως σε θέματα όπου η νομική υπηρεσία έχει ήδη εκφράσει την απόψή της. Τέλος, κάτι χρήσιμο για μία μόνιμη συνεργασία που μπορούμε να προσφέρουμε στα μέλη της Επιτροπής Ελευθεριών είναι η εξέλιξη ε, του ε, εθνικού δικαίου εις ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μπορούν όλοι να γνωρίζουν τις γενικές αρχές στις οποίες βασίζεται το ποινικό δικαίου και για να απαντήσω εις τα ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή Επιτροπή θα σας πω ότι η εμπειρία του παρελθόντος μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια σαφή ιδέα της μεθοδολογίας που πρέπει να εφαρμόσουμε για να υπάρχει πιο αποτελεσματική ε, χρήση. Χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση και αυτό προϋποθέτει ότι τα κράτη θα μπορούν συνέχεια να παρακολουθούν την νομική διαδικασία σε κάθε σημείο και ότι η επαγγελματική επιμόρφωση είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε και μία μόνιμη συνεργασία με τα ε, υπόλοιπα θεσμικά όργανα θα μπορέσει να εξασφαλίσει εξαιρετικής ποιότητος υπηρεσίες ε, και ε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήματα. Ναι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Δεν έχουμε χρόνο και οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν. Και αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια, σας παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. Και κατόπιν θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Παρακαλώ σε σχέση με την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα. Εμείς, ε, οι Ευρωβουλευτές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία όταν ε, μιλάμε για νομοθεσία πρόληψης και κυρίως για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εδώ πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί υπογράφουμε συμφωνίες με άλλες χώρες, με τις Πολιτείες λόγου χάρη, όπου αυτό που θέτουν δεν είναι νομοθετημένο στην, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένε φορές ούτε καν στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να αξιολογήσουμε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα. Εγώ τώρα δεν είμαι εισηγήτρια, αλλά είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό PNR και φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή των ατόμων. Υπάρχει αυτό το αγαθό, αλλά αυτό περιορίζεται γιατί έχουμε και την συνιστόσα της ασφάλειας. Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι τα αδικήματα που αιτιολογούν μια παρόμοια νομοθεσία γιατί μιλάμε για πάρα πολύ διαφορετικά δικήματα που θα μπορούσαν ε, να ληφθούν υπόψη, όπως ε, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα ή σοβαρά εγκλήματα, όπως τα αποκαλούμε. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ενολογικότητα εδώ, καθώς ε, οι πηγές των πληροφοριών είναι αστυνομικές και δεν μας αναφέρουν ρητός αυτέ τι πληροφορίε. Έχουμε πάρα πολλέ δυσκολίε λοιπόν στο θέμα αυτό και στρέφουμε στην Κομισιόν γιατί υπάρχει πρώτη οδηγία επιτάπητο. Έτσι λοιπόν, ίσω αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δουν μια ομάδα, να τα δει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να γίνει εξελόξη. Γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία στα κρατη και η ευρωπαϊκή νομοθεσία ουσιαστικά επιβάλλεται να ληφθεί επειδή υπάρχουν διεθνεί συμβάσει. Και κοιτάξτε, η πρόληψη στους ποινικού κώδικες καθυστερεί πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Να ευχαριστώ, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία μας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι αυτό το εγχειρήμα θα είναι η αρχή όχι το τέλος μια πολύ πιο αυστηρού αξιολόγηση για την αδερφή πληροφοριών μεταξύ των τριών ε, οργάνων ε, και σημείωσε και την επίνομικη υπηρεσία ε, του Κοινοβουλίου ότι δεν υπάρχει επαρκή προσωπικό και πρέπει τώρα να μεγιστοποιήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών των οργάνων μας. Γίνεται πολύ μεγάλη εξέταση στο ιστορικό της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι πιο προδραστικό στο να εμπλέξει και το Κοινοβούλιο. Και επίσης ε, υπήρχε και μια δηλώση πρακτικών του Συμβουλίου όταν ε, θετήθηκαν ε, αυτές, αυτά τα συμπεράσματα για τις πρότυπες διατάξεις. Υπήρξε μια δήλωση της Κομισιόν στα πρακτικά ότι θεωρεί η Κομισιόν τις διατάξεις αυτές ε, μια προημή και περιορισμένη ερμηνεία του άρθρου 83. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ αρχίζουμε τελικά να σκάβουμε και να αναδύονται κάποιες από τις εντάσεις σε όλα αυτά. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς κρυβόταν πίσω από αυτή τη δήλωση της Κομισιόν και Σημείωσε ότι είπε και ο κύριο Στροπόλσκι τη Πολωνική προεδρία. Ε, είπε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να πάνε παραπέρα στο εθνικό δίκαιο. Αναφέρθηκε σε συμπέρασμα του Συμβουλίου από το Παλαιθόν. Νομίζω ότι αναφερθόταν στι ποινέ. αλλά ξέρω με τον κύριο Νιτσέ να αναφέρεται στην δυνατότητα αν ποινικοποιείται η πρόθεση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το κράτος μέλος ε, δεν μπορεί να ποινικοποιήσει την αμέλεια. Και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και μάλιστα, χθες το βράδυ, ε, ουσιαστικά ε, Νομίζω ότι ε, θα κάνω μια προσφυγή στον ε, Βουλή των Λόρδων ε, για τις ποινικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και μια νέα οδηγία που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη ότι η δίωξη δεν εξαρτάται από το να υπάρχει καταγγελία από το θύμα και παραδείγματος χάρη μπορεί να αποφευκτεί η δίωξη αν αναγκαστεί το θύμα να καταθέσει. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μέτρο ουσιαστικού δικαίου που νομίζω ότι έχει αποτελέσμα spillover σε δίκο οικονομικές πτυχές. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ακρόαση αυτή, αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ε, μεταξύ των τριών οργάνων. Ευχαριστώ. Και ωραία. Ξέρω ότι μας λείπει ο χρόνος, αλλά τι να κάνουμε λοιπόν. Ο κύριος Πρίμπερ είναι εδώ και θέλει και αυτός να μιλήσει. μετά θα μιλήσουν και οι άλλοι και οι άλλοι όλοι θα μιλήσουν εδώ. Γι' αυτό μας λείπει ο χρόνος. Λοιπόν, κύριε Πρίμπη πρώτα και μετά το Συμβούλιο και μετά το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μόνο να σας πω μερικά, μερικές πληροφορίες στη χρήσιμη αυτή συζήτηση. Πρώτον, δύο χρόνια μετά την έναρξη της συνθήκης της Λισαβόνας δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα νομοθεσίας για το θέμα που μας αφορά. Δηλαδή, από τις γενικές συζητήσεις και αναλύσεις που κάνουμε πρέπει να κινηθούμε προς την λήψη μαθημάτων από τις πρώτες σχετικές νομοθεσίες που είναι η οδηγία για τη δουλεμπορία και την κατάχρηση των παιδών. Υπάρχουν καταστάσεις όπου παρά τις κατανοητές αμφιβολίες των χωρών μελών για να δεχτούν παρέμβαση σε ενωσιακό ποινικό δίκαιο, Υπάρχει και η πολιτική θέληση να γίνει κάτι τέτοιο όπως φάνηκε από την οδηγία για το δουλεμπόριο. Τι μαθήματα λοιπόν πήραμε από αυτή την νομοθεσία. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχουν τομείς όπου τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν αλλά θέλουμε η νομοθεσία να είναι πολύ υψηλού επίπεδου, αλλιώς θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες επικρίσεις. Επίσης δεν πρέπει να βάζουμε τέτοιου είδους νομοθετικές ρήτρε που δεν είναι ακριβώς ποινικό δίκαιο αλλά συνδέεται με αυτό σε όλα τα θέματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι πολύ σωστές και χρήσιμες, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην δεσμευτούμε χωρίς να χρειάζεται απολύτως κάτι τέτοιο. Αυτό. Ο Στρόφκης. Ευχαριστώ. να απαντήσω στην κυρία Ραμέρο Ναι, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για τα ίδια εγκλήματα, όντως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθεί, να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό γρήγορα. Αντί όμως να ζητήσουμε εναρμόνιση των ορισμών, Ίσως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, δηλαδή να συμπληρωθούν οι συμφωνίες με ασφαλιστικές ρήτρε. Θα ήταν και αυτός ένας τρόπος να υπάρξει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια αντί να ζητηθεί πλήρης εναρμόνιση. Για τις θεσμικές εντάσεις που παρατηρήθηκαν δεν οφείλονται νομίζω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από εκείνες και να θεωρήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου ως πολύτιμη συμβολή και βάση περαιτέρω ανάλυσης. Και οι τελευταίες δηλώσεις της Κομισιόν για τις χειραγωγήσεις της αγοράς δεν λένε τίποτα διαφορετικό βασίζονται σε αυτές τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές. Και εγώ σύντομος. Εμείς θα θέλαμε πολύ στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς και όργανα. Και πήραμε πολλά μαθήματα εμείς γιατί συνεχίζουμε την ανάλυση μας και σκεφτόμαστε μήπως πρέπει και μπορεί να γίνει μια πολύ πιο ενεργή παρέμβαση της νομικής υπηρεσίας, να πληροφορεί δηλαδή τακτικά για τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, παραδείγματος χάρη, στο ερώτημα της κυρίας Ρομέρο Λόπες για την πρόληψη των εγκλημάτων, ήδη στη νομική υπηρεσία κάνουμε μια εσωτερική συζήτηση της πρακτικότερης δυνατής εφαρμογής του άρθρου 84 για την πρόληψη του εγκλήματος. Μέχρι τώρα δεν έχει αναλυφθεί κανένα μέτρο με βάση το άρθρο αυτό και ίσως θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε και αυτό σε μελλοντικέ ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών μα και του Κοινοβουλίου, καθώ και των υπηρεσιών μα και του Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Αυτό χρειάζεται ολόκληρη άλλη ακρόαση όπως καταλαβαίνετε. Τώρα ο κύριος Ντε να συνοψίσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους ε, διερμηνείς Δεν θα με κρηγορήσω, δεν θα σας πω τι έμαθα σήμερα το πρωί. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που και για μένα ήταν καινούρια, κυρίως το θέμα της αξιολόγησης, το στοιχείο της αξιολόγησης. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ ε, προσεκτική προετοιμασία της νέας νομοθεσίας, ναι μένω, αλλά πρέπει να εξετάζουμε και πολύ προσεκτικά όσα ήδη χρησιμοποιούμε. Εγώ θέλω να πω στους ε, σκιώδεις ότι θα εκπονήσω ένα έγγραφο που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ακούσαμε σήμερα το πρωί και θα βασίζεται ε, στο διάγραμμα που γνωρίζουν ήδη οι σκιώδεις και έχω εκπονήσει νωρίτερα φέτος και νομίζω ότι είναι καλό να διαβουλευτούμε και με ορισμένους ε, ε, με του εμπειρογνώμονε που τον σήμερα το πρωί λόγου χάρη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι περί τα μέσα τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε το σχέδιο τη έκθεση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κοινή δουλειά μα και ανυπομονώ. Και φυσικά συμφωνώ ότι όπω είπε η κυρία Λέτβερ θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.